Colleagues, good morning. Please be seated. Uh, Καλημέρα συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. ξεκινήσουμε με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά και στο ίντερνετ. Διαθέτουμε διερμηνία για τις γλώσσες που μιλούν οι, τα μέλη της Επιτροπής. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 6 Φεβρουαρίου 2017. Έχετε δυνατότητα να υποβάλλετε παρατηρήσεις στα πρακτικά μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Σε διαφορετική περίπτωση τα πρακτικά θεωρείται ότι εγκρίνονται. Ας εγκρίνουμε τώρα την ημερήσια διάταξη. Δεν έχει υποβληθεί κάποια ένσταση, κάποια παρατήρηση. Επομένω, εγκρίνεται και η ημερήσια διάταξη. Το τέταρτο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας θα το εξετάσουμε από με, τα, τα, μέλη της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, της ΔΕΒΕ και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας, τον κύριο Γκέρατς συζήτηση ε, σήμερα θα εστιάσει στην κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό και βεβαίω η αναπτυξιακή βοήθεια για την περιοχή αυτή είναι πολύ σημαντική. Εξού και η συνεδρίασή μα από κοινού με την Επιτροπή ΤΕΒΕ. Το απόγευμα θα έχουμε μια δημόσια κρόαση για την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στην Ασία και τον Ειρηνικό στη θάλασσα της Ανατολικής και Νότιας Κίνας και στο τέλος θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις της Ηνωμένες Ε, έχω μία ε, ανακοίνωση να σας κάνω. Θα πρέπει να κλείσουμε την ε, συζήτηση ε, 10 παρα 10 έτσι ώστε να ε, παρευρεθούμε και εμείς στην εκδήλωση που θα γίνει που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κ. Σταγιάννη για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες ε, στις 22 Μαρτίου πέρυσι. για να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση μέχρι εκείνη την ε, ώρα, τη συζήτηση αυτού του σημείου δηλαδή, θα προσπαθήσω να δω πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για το Κονγκό και είτε θα κλείσουμε αυτό το σημείο της της διάταξης πριν τις 10 παρα 10 και θα επαναλάβουμε τις συνεδρίες στις 10.30 ε, ε, συζητώντας για την πολιτική ασφαλείας και άμυνας ε, και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, δηλαδή το επόμενο θέμα, ή εναλλακτικά θα επιστρέψουμε αμέσως και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το Ανατολικό Κόγκο, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση. Θα δώσω αμέσως τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρενς για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. και μετά στους ομιλητές, τους οποίους και θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Ο κ. Κάρπεντερ, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος για την Κεντρική Αφρική, ε, συντονιστής για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και δίνω το λόγο αμέσως στον κ. Γκέρενς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, διοργάνωση από κοινού με την Επιτροπή μας αυτής της συνεδρίασης, έτσι ώστε να συζητήσουμε για τα ζητήματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είναι και το αντικείμενο της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για τους συναδέλφους εκείνους ε, μάλλον θα, θα κάνω τι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει για του συναδέλφους, ο κ. που είναι αρκετά πρωινή για να παρευρίσκονται αργότερα. Ε, ευχαριστούμε κύριε Γκέρεν. Να σα υπενθυμίσω ότι ότι ο λόγο που συζητούμε αυτό το θέμα και το έχουμε στην ημερησία μα διάταξη είναι επειδή πρόκειται να διοργανώσουμε μια αποστολή στο Ανατολικό Κονγκό στην οποία θα συμμετάσχουν και τρία μέλη της Επιτροπής και υποφαινόμενοι και θέλαμε να έχουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο κύριε Κάρπεντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Θα αρχίσω, αν μου επιτρέπετε, γιατί αρχικά η πρόθεση ήταν να έρθει και από το ΝΟΙΕ κάποιο ομιλητή. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Εμεί στη διεθνή κοινότητα εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό για την ενημέρωσή μα για την ε, κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό στο έργο των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ. Πριν από δέκα μέρες, δύο μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων και τέσσερις ε, Κογκολέζοι εξαφανίστηκαν στο κεντρικό Κασάι και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ευθύ εξ αρχής την αλληλεγγύη μας με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να εκφράσουμε θερμές ευχές για την ασφαλή επιστροφή των εμπειρογνωμόνων ε, και να εκφράσουμε και την εκτίμησή μας για το έργο τους. Είμαι ευγνώμων για τη σημερινή πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της Επιτροπής σας και της Επιτροπής ΔΕΒΕ για την, ε, ε, την ανατολική περιοχή του Κονγκό. Ε, αυτό έχει να κάνει και με τις ε, προκλήσεις που υπάρχουν και έχουν προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα, ιδιαίτερα επειδή είναι εκλογική χρονιά φέτος, ε, μια χρονιά κατά την οποία η χώρα θα κάνει ένα σημαντικό βήμα και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της σταθεροποίησης. Θέλω να πω δύο λόγια για την κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό όπως τη βλέπουμε και να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εστιάσουμε σε ένα σημαντικό θέμα σήμερα το οποίο είναι η επαναδιαπραγμάτευση της εντολής για το Μονούσκο, δηλαδή την παρουσία του ΟΗΕ στο Ανατολικό Κονγκό. Καταρχήν, ε, αν έχετε διαβάσει την πρόσφατη έκθεση των εμπειρογνωμών και παρακολουθείτε τις εξελίξεις στη χώρα αυτή, δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακόμα αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα από τις ένοπλες ομάδες. Ε, και στο Κίβου, ε, η VADF, για παράδειγμα, η FDLR και ενδεχομένως και μια ε, ανάδυση πάλι και άλλων ομάδων που λειτουργούν γενικότερα στο Ανατολικό Κονγκό, δηλαδή ο, ο στρατός της αντίστασης, ε, ένοπλες ε, ομάδες τοπικές. Ε, είναι πολλά τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αρκεί να πούμε αυτή τη στιγμή ότι στην περίπτωση του FDLR ε, αποδυναμώθηκε το 2016 και διασπάστηκε, αλλά είναι ακόμα μια μεγάλη απειλή παρά την αποσταθεροποίηση. Η ADF ιδιαίτερα και όπως είπαν και οι εμπειρογνώμονες, ε, αυτοί συνεχίζουν να στρατολογούν, να εκπαιδεύουν και να λειτουργούν ενεργά, προκαλώντας μεγάλη ανασφάλεια στις ε, περιοχές όπου εξακολουθεί να δραστηριοποιείται η ομάδα αυτή. Το πρόβλημα των ενόπλων ομάδων και η ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν δείχνει μία μια ε, αποτυχία σε, άλλες, ε, σε, σε άλλους τομείς. Ε, δηλαδή να υπάρξουν διαδικασίες καινούργιες, δηλαδή αυτές που απορρέουν από τις διακηρύξεις του Ναϊρόμπι που σηματοδοτούν το τέλος της εξέγερσης και το άλλο είναι το πλαίσιο της συνεργασίας για την ειρήνη και της, ε, που ε, ενέχει πολλές δεσμεύσεις ε, για την μακροχρόνια ανάπτυξη και σταθεροποίηση του Ανατολικού Κονγκό. Αυτό καθ' αυτό και η έλλειψη πολιτικής δράσης, αν θέλετε, δείχνουν κάποιοι κάποιες, ε, κάποια σοβαρά προβλήματα σε εθνικό επίπεδο, στις μεγάλες λίμνες. Ε, δύο που δεν θα σας εκπλήξουν είναι η κρίση στο Μπουρούντι, που εξακολουθεί να είναι πρόκληση για την περιοχή και το δεύτερο πρόβλημα είναι βέβαια η πολιτική κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό που εστιάζεται στην προετοιμασία των εκλογών που ελπίζομαι ότι θα μπορέσουν να διεξαχθούν το 2017. Έχουμε λοιπόν μια επισφαλή κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό. Ακόμα δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για ασφαλείς νησίδες σταθερότητα. Να προσθέσουμε εδώ σκεπτόμενοι και την ικανότητα του Μονούσκο και ε, του επίσημου στρατού να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το γεγονός ότι έχουμε νέα σημεία πίεση στη χώρα είτε στο Κασάι ε, λόγω της εξέγερσης ε, ε, εκεί και των νέων προκλήσεων από τις ένοπλες ομάδες αλλά και άλλες πιέσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέχρι τις εκλογές και με τη διαδικασία καταγραφής και τις πολιτικές διαδικασίες γενικότερα θα είναι δύσκολο να δούμε πού και να προβλέψουμε πού θα δημιουργηθούν αιστείες, εστίες ανασφάλειας που δεν θα έχουν να κάνουν με τις παραδοσιακές εξελίξεις που ξέραμε. Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο Κονγκό και στο Ανατολικό με καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό αναφέρεται στην έκθεση των εμπειρογνωμών και στην έκθεση ε, του Γενικού Γραμματέα στο Συμβουλίο Ασφαλείας. Φαίνεται ότι οι καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυξάνονται και δυστυχώς τονίζεται και το μεγάλο ποσοστό καταχρήσεων από κρατικούς αξιωματούχους. Έχουμε θέματα και στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Ε, πολλοί είναι οι εκτοπισμένοι στο Κονγκό. Εξακολουθήσει η κατάσταση αυτή να υπάρχει μέχρι το τέλος του 2016. Ε, μετά από αυτή τη σύντομη περιγραφή θα ήθελα να περάσω τώρα στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο εύκολο για να αρχίσω, γιατί είναι η επίσημη θέση μας ε, πρόσφατα, το, στα συμπεράσματα του Μαρτίου του Συμβουλίου. Προφανώς συνεχίζουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση στο Κονγκό γενικότερα. Καλωσορίζουμε την πολιτική συμφωνία που επετέχθη στη 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά την ε, ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας αυτής ε, μέσα από το αρανσμό παρτικιουλία, δηλαδή τις ειδικές, τους ειδικούς διακανονισμούς για τη συμφωνία που εξακολουθούν να ε, εφαρμόζονται. Εκφράζουμε την επιθυμία μας για ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας και ειδικότερα για η προεδρική πλειοψηφία να παίξει το ρόλο της με στόχο να γίνουν οι εκλογές πριν από το τέλος του 2017. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το έργο της διάσκεψης των καθολικών επισκόπων που ήταν πάρα πολύ σημαντική για να υπάρξει πολιτική συνένεση τότε που ε, έγινε. Τονίζω ότι για μας τώρα, και αυτό αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ε, δεν πρόκειται μόνο για κρίση ασφάλειας ε, στο Ανατολικό Κονγκό. Από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε πολυδιάστατη, πολυδιάστατη κρίση ε, και θεσμική και κοινωνικο-οικονομική πέρα από θέματα ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σχετικά και αλληλένδετα όταν εξετάζουμε τις προοπτικές ασφαλείας στη χώρα το 2017. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανανέωση της εντολής Μονούσκο. Νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, επικέντρωσε καταρχήν στην ανάγκη η αποστολή να έχει τα μέσα που χρειάζεται, ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα να μπορεί να συνεχίσει να πληρεί το ρόλο της προστατεύοντας τον πληθυσμό και βέβαια ετοιμάζοντα και τις εκλογές γιατί το Μονούσκο παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά επίπεδα. Συνεχίζουμε να καταδικάζουμε τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιοι θα γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε επιβάλει κυρώσεις κατά ορισμένων ατόμων σε σχέση με άσκηση βίας πέρσι το φθινόπωρο. Ε, εκφράσαμε την ετοιμότητά μας να εφαρμόσουμε νέες κυρώσεις ε, αν χρειαστεί ε, για τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παρακόλληση των πολιτικών διαδικασιών συνεχίζουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας για την ανθρωπιστική κατάσταση και σημειώνουμε ειδικότερα ανησυχίες στο Ανατολικό Κονγκό, στο Κιβούς, στην τανκανίκα και δεν πρέπει να παραλείψω και τον Βορρά όπου συνεχίζεται η κατάσταση στο Καράμπα Πάρκ και τα σώματα αντίστασης. Υπενθυμίζομαι τις δεσμεύσεις της διακήρυξης του Ναϊρόμπι και αυτές που απορρέουν από το πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης, που είναι για μας ο κεντρικός πυλώνας, αν θέλετε όταν χειριζόμεθα το θέμα του M23 αλλά και άλλα θέματα. Για να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, θα πω δύο λόγια για το Μουνούσκο. Ε, πρώτα όμως να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει οικονομικά πολλές διαδικασίες που είναι σημαντικές για το Ανατολικό Κονγκό. Τονίζω ένα πρόγραμμα σταθερότητας, αν θέλετε, που έχει να κάνει με ένα μηχανισμό για την σταθερότητα και την ειρήνη, τη στρατιωτική δικαιοσύνη, η οποία είναι πολύ σημαντική, αν θέλουμε να αποφύγουμε την ατιμορρησία ε, των ενόπλων δυνάμεων. Να τονίσω ακόμη ότι εξακολουθούμε να, ε, κάνουμε, να συμβάλλουμε στις διορθωτικές αλλαγές στο στρατό. Ε, ολοκληρώσαμε την αποστολή μας η πριν από ένα χρόνο, αλλά εξακολουθούμε να εργαζόμεθα με αναπτυξιακά κονδύλια για το στρατό, για τον εξυγχρονισμό της διοίκησης και τη λογοδοσία, όπως θα την ονόμαζα, των ενόπλων δυνάμεων ενώπιον του Κοινοβουλίου αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Για το Μονούσκο η συζήτηση για την εντολή είναι κέρια σημασίας. Προφανώς αυτό είναι θέμα που θα αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας σε ό,τι αφορά τις προθέσεις που θα έχει δηλαδή, αλλά η εντολή και τα μέσα που αποδίδονται στο Μονούσκο χρειάζονται για να παίξει το ρόλο του στα πλαίσια της προστασίας αλλά και των εκλογών. Η συζήτηση στη Νέα Υόρκη σε σχέση με την Συμφωνία για την Τελική Εντολή αναγνωρίζει όλα τα κέρια ζητήματα αλλά και τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν το Ανατολικό Κονγκό ε, θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν και πρέπει να παρακολουθούνται είναι Πρώτον, η ταχεία ολοκλήρωση του αρασμό των παρτικούλια για τη συμφωνία. Επίσης θα πρέπει να ε, καλυφθούν ε, στην εντολή Μονούσκο ικανοποιητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβάνοντας ε, διώξεις από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων τα, οι εθνικοί θεσμοί στο Κονγκό θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, για παράδειγμα κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα αναθεωρήσει τον εκλογικό νόμο, ώστε να ε, τηρηθούν οι προθεσμίες για τις ε, ένοπλες ομάδες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, σεβαστούν τα, τις δεσμεύσεις της συμφωνίας και να σεβαστούν και τις κυρώσεις του ΟΗΕ που αφορούν τις ένοπλες ομάδες και βέβαια ε, τα ενεχόμενα μέρη της διακήρυξης του νερό πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Μας ενδιαφέρει προφανώς ε, η δραστηριότητα των ε, στρατευμάτων και των ενόπλων ομάδων Ε, ε, κλείνω εδώ, θα ήμουν ευτυχής να απαντήσω σε ερωτήσεις. Να πω όμως ότι για μας το 2017 είναι ένα έτος όπου η πολιτική βούληση όλων θα τεθεί σε δοκιμασία, όλων των ενεχομένων μέσα στη χώρα, οι δυνάμεις που δρούν προς το εθνικό συμφέρον για να επιτύχουν ε, εκλογές ικανοποιητικές, αλλά θα δοκιμαστεί και η πολιτική βούληση της διεθνούς κοινότητας που θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα αυτή διατηρώντας ε, τα επίπεδα στήριξης του έργου των Ηνωμένων Εθνών ε, βοηθώντας το λαό του Κονγκό να επιτύχει το στόχο που αξίζει να επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Κάρπεντερ, για την πολύ εκτεταμένη εισαγωγή σας. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα, θέλαμε να καταλήξουμε σε μία δήλωση που θα εκφράζει την αλληλεγγύη μας προς την ομάδα εμπειρογνωμόνων και την εξαφάνιση των μελών, κάποιων μελών της ομάδας, η οποία προσπαθεί να στηρίξει το Κονγκό. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προετοιμασία της, την της αποστολής που θα πάει στο Ανατολικό Κονγκό. Μέσα σε τέτοιες ε, συνθήκες, σε μια τέτοια συγκυρία, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε τώρα. Μια και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να σταθεροποιήσουμε τη χώρα. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε όλες αυτές τις επιλογές που παρουσίασε ο κύριος Κάρπεντερ μέσα στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. μετά την ε, επιτυχή αρχική εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεξαχθούν εκλογές. Εκλογές μέσα στο 2017 στο Κονγκό. Ο κύριος Γκάλερ. Φαντάζομαι θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχα ένα ραντεβού με τον γιατρό. Σας ευχαριστούμε για την ε, ενημέρωση που μας κάνατε για την κατάσταση στη χώρα. Η ερώτηση που θέτω και στον εαυτό μου εδώ και καιρό, όχι μόνο σήμερα, είναι ωραία. Μη είμαστε ενημερωμένοι. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει από πλευράς μας και νομίζω ότι βοηθάμε τις αρμόδιες αρχές, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση παραμένει η ίδια. Φυσικά στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΟΗΕ, αλλά για να υπάρξει πραγματική αλλαγή στη χώρα, δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να στείλουμε μια πραγματική αποστολή στη χώρα, κάτι ουσιαστικό. Γιατί όπως βλέπετε σε αυτή την περιοχή των μεγάλων λιμνών, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει πραγματική διοίκηση, σοβαρή διοίκηση, η οποία θα βοηθήσει τον πληθυσμό. Και όλα αυτά τα ελλείμματα τα οποία περι, ε, ε, περιγράφουμε, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Το μόνο πράγμα που θα έκανε τη διαφορά θα ήταν κάτι τέτοιο. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι, να στηρίξουμε το έργο του ΟΗΕ. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική βούληση στη χώρα. Και δεν το κρίνω καν, δεν το κριτικάρω καν. Ίσως έχουν άλλες προτεραιότητες όσο τραγικό και αν είναι. Τι να πω, μου προξενεί απόγνωση, απεσιοδοξία. Άκουσα αυτή τη ρεαλιστική περιγραφή σας, αλλά πώς μπορούμε με αυτά τα δεδομένα εμείς να κάνουμε τη διαφορά. Συμφωνώ απόλυτα. Πριν από 10 χρόνια είχαμε μια μεγαλύτερη βούληση να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε τη χώρα. Κυρία Βάουτμαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας επιτρέπετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Ήταν από το 2014 και παραμένει ακόμα ανησυχητική. Ολόκληρα χωριά καίγονται, έχουν καεί. Άνθρωποι δολοφονούνται, παιδιά στρατολογούνται ως στρατιώτες. Υπάρχει και μία σεξουαλική γενοκτονία. Τα θύματα απαξιώνονται, στερούνται την αξιοπρέπειά τους. Ε, το θέμα συζητιέται και στον ΟΗΕ. Το θέμα είναι τεράστιο όμω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η κατάσταση. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Κοιτάξτε τα νούμερα. Το 2014 ε, δολοφονήθηκαν 700 με 1000, ε, 1.300 άτομα. Και άνθρωποι εξαφανίζονταν κτλ. Αυτές είναι μόνο εκτιμήσεις. Τα πραγματικά νούμερα ίσως είναι πολύ μεγαλύτερα. Τώρα έχουμε τη Μονέσκου επιτόπου. Νομίζω ότι η εντολή της πρέπει να ενισχυθεί. Και επίσης πρέπει να παρακολουθούμε τι κάνει η UNESCO. Η UNESCO. Γιατί μερικές φορές ακούμε ιστορίες ότι η UNESCO παίζει το ρόλο του παρατηρητή και απλώς βλέπει τις φρικαλαιότητες που συμβαίνουν. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η βία θα αυξηθεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, και να δούμε τι κάνει η Μονούσκο. Ξέρετε ότι υπάρχει μια έκθεση που ετοιμάζουμε Υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλά θύματα και η ομάδα αυτή η οποία ασχολείται με, την κατάσταση των θυμάτων προσπαθεί να, δώσει, ε, να βάλει όνομα στα θύματα για να μην είναι, και να μην παραμείνουν ανώνυμα. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη δήλωση ότι αυτό που θέλουμε είναι να γίνει μια ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή ε, για να χυθεί απλό το φως στο ποιοι είναι οι Γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, όχι απλώς ε, δολοφονούνται άνθρωποι, όχι απλώς υπάρχουν θύματα, αλλά λόγω της ανωνυμίας γίνονται θύματα δεύτερη φορά. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να αποκαλυφθούν. Και σε ό,τι αφορά γενικά το Κονγκό, ο λαός είναι θύμα, αλλά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, θα πρέπει να τη ασκήσουμε πίεση, ούτω ώστε να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κογκολέζικο στρατό, πολύ συχνά εμπλέκεται σε πράξει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι κάνει η Ευρώπη, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί. Πώ μπορούμε να δώσουμε περισσότερε εξουσίε στην Επιτροπή και εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε, μπορούμε να στείλουμε παρατηρητές, τι ρόλο θα μπορούσαμε να παίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε τις περιπτώσεις μαζικής παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει ατιμορρησία ούτε στο Κονγκό, αλλά ούτε σε άλλες αφρικανικές χώρες. Ευχαριστώ. Θέλω να στηρίξω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι καταρχάς, κυρίως ε, τα όσα είπε ο κύριος Γκάλερ. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματική παρουσία στη χώρα αυτή. Μιλήσαμε για 10 ε, για τους θανάτους στη Συρία, ενώ στην, την περιοχή των μεγάλων λιμνών θα έχουμε, έχουμε ήδη 10.000 θύματα. Ε, όσο δεν θα έχουμε ένα πραγματικό στρατό που να κάνει επιθέσεις δηλαδή, και δεν μιλάω για τη Μονούσκο η οποία είναι παρατηρητής απλώς, παρατηρεί τις φρικαλαιότητες, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη. Εγώ ε, πήγα σε αυτή τη χώρα υπό την αιγίδα του στρατηγού Μαρόλ με το Ζαϊντίν Γκομά εν συνεχεία. Ξέρω πολύ καλά την ιστορία του Καμπίλα, Ξέρω πολύ καλά τις επιχειρήσεις που κάνει ξένες δυνάμεις. Στην πραγματικότητα ετοιμάστηκε μια λαιλασία. Ε, την ενορχίστρωσαν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι παρόντες ε, στο, στη Ρουάντα και που εξάγουν κοβάλτιο Θα πρέπει λοιπόν από τη μία να έχουμε παρουσία επιτόπου, να κάνουμε μια σοβαρή ανάλυση για το ρόλο των ε, ξένων δυνάμεων και των υπηρεσιών τους, που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο, άμεσα εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο. Εγώ ε, ήμουνα ένας από τους ε, συντάκτες ε, μιας έκθεσης για τους πολέμους για την έκκληση για πόλεμο, έτσι λεγόταν αυτή η έκθεση. Αλλά εκεί ακριβώς λέγαμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια, ε, ένα θύλακα ελεύθερο ας πούμε, όπου θα πηγαίνουμε και θα διώχνουμε, θα εξαφανίζουμε τους αντάρτες. Όλα αυτά επίσης πρέπει να τα δούμε σε σχέση με το ρόλο που έχει παίξει η Ρουάντα η Ρουάντα είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Καγκαμέ παίζει ωραία το παιχνίδι του. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και τον πραγματικό ρόλο της Ρουάντα στην αποσταθεροποίηση του Κονγκό ε, που τη βοήθησαν και οι ξένες δυνάμεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Συζητούμε την κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό, την Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και βλέπω ότι δεν ζητούν το λόγο άλλοι συνάδελφοι, επομένω κύριε Γκέρενς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, δεν είναι πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα αυτό. Τα τελευταίους δέκα μήνες έχουμε κρίνει μάλιστα και δύο ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία αφορούσαν αφενός στην καθυστέρηση στις εκλογές το οποίο μας ανησυχεί όταν διαπιστώνουμε ότι ένας ε, πρόεδρος ε, αυτής της χώρας, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να ανανεώσει τη θητεία του σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, ε, παρόλα αυτά προσπαθεί να παραμείνει. Το δεύτερο σημείο. Αυτή, αυτό το τελευταίο ήταν μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, έρχομαι στις, παρα, στις παρατηρήσεις του κυρίου Κάρπεντερ. Ε, κάποιος ο οποίος εργαζόταν στο Ανατολικό Κόγκο μας είπε ότι αποφάσισε, ε, σκεφτόταν μάλλον να σταματήσει να εργάζεται γιατί ήταν πλέον αδύνατον και το συζητούσε με τη γυναίκα του και είπε ότι όχι, παρόλα αυτά θα θέλω να συνεχίσω την, ε, δουλειά μου εκεί γιατί δεν μπορώ να προδώσω ανθρώπους όπως αυτούς που είχα γνωρίσει μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία ε, η οποία είχε ένα παιδί από βιασμό για να σας δώσω μια εικόνα για τις ιστορίες που ακούει κανείς από αυτήν την περιοχή είπατε ότι χρειάζεται να κάνουμε μια διάγνωση. Είναι η συνηθισμένη κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. όπου έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος εξελέγει πρόεδρος σε μια διεφθαρμένη χώρα και γιατί είναι διεφθαρμένη η χώρα, γιατί η δημόσια πάλι είναι διεφθαρμένοι. Γιατί είναι διεφθαρμένη εκείνη, γιατί δεν ε, έχουμε χρήματα στον προπολογισμό για να ε, δώσουμε μισθού. Και γιατί είναι έτσι η κατάσταση του προπολογισμού, γιατί η κατάσταση τη χώρα είναι ε, ότι η διαφθορά βασιλεύει. Γι' αυτό το λόγο κανένα ξένο επενδυτή, ένα Γάλλο για παράδειγμα, δεν πρόκειται να επενδύσει. Και ο προπολογισμό τη χώρα παραμένει σε άσχημη κατάσταση, τα έσοδα τη. Επομένω, έχουμε ένα φαυλο κύκλο τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο που ανέφεραν και πολλοί από τους προσλαλήσαντες είναι η ενίσχυση του ρόλου των, της, ε, των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι ώστε να καλύψουμε το κενό εξουσίας που υπάρχει. Και γιατί είναι, υπάρχει αυτό το κενό εξουσίας εξαιτίας της διαφθοράς και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων, όχι μόνο ε, των κρατικών φορέων, αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν για να ε, ενισχυθεί η τοπική διακυβέρνηση. Και έτσι ώστε από την τοπική διακυβέρνηση σιγά σιγά να χτιστεί ένα κράτος, να φτάσουμε στην ε, κρατική διακυβέρνηση. Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας. Επομένως, είναι ορθό που επαναλαμβάνουμε ε, συνεχώς ότι η παρουσία της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να ενισχυθεί. Τρίτον, ε, κύριε Κάρπεντερ είπατε ότι τα κοντήλια που είναι διαθέσιμα τα χρησιμοποιείται επίσης και για την εκπαίδευση του στρατού και πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο. Στη, τα, τα πρώτα χρόνια της, μετά τον πόλεμο, δηλαδή πριν 12 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε με τη χρηματοδότηση του ε, χρηματοδοτικού εργαλείου για την ειρήνη στην Αφρική. Είχαμε δώσει χρήματα με κατά κύριο λόγο ε, για αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και το έγγραφο Responsibility to Protect, η ευθύνη για να προστατεύουμε τους ανθρώπους που αναφέρεται σε περιοχές της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένες και της, του, του, του, περιοχής για την οποία μιλάμε, ε, για την, κατάσταση στο Ανατολικό Κονγκό και στο οποίο αναφέρεται και παριγράφεται πώς η, το, τα προβλήματα ασφαλείας ε, οδηγούν τελικά στο να μην μπορεί να αξιοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια. ευχαριστώ. Κύριε Κάρπεντερ, Έχετε περίπου 10 λεπτά για να απαντήσετε. Και μετά θα ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και σας παρακαλώ να ε, κατεβούμε όλοι μαζί κάτω για το θέμα που είπαμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Να αρχίσω ίσως από την τελευταία παρατήρηση, ή την πρώτη τελευταία μάλλον του κυρίου Γκέρνς γιατί είναι ενδιαφέρουσα, έχει να κάνει με μια χαρτογράφηση, αν θέλετε, των κρατικών και μη κρατικών φορέων που παίζουν ρόλο. Θα προσθέσω εδώ και μια χαρτογράφηση των ε, νόμιμων παικτών, κρατικών και μη. Ε, εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση μεταξύ ευθυνών μας βράχη και μακροχρόνιων. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρέπει να πούμε ότι ε, οι μακροχρόνιες ε, ε, ευθύνες είναι πολλές και οι εκλογές θα παίξουν το ρόλο του καταλήτη εδώ. μακροπρόθεσμα θέλω να δουλέψουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, για τα δημόσια οικονομικά, για τον τομέα της υγείας στο Κονγκό και τίποτα από αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς αποτελεσματικό και διαρθρωμένο διάλογο με έναν νόμιμο, νομιμοποιημένο δηλαδή ε, συνομιλητή. Αυτό είναι δύσκολο σήμερα και γι' αυτό μεταξύ άλλων ε, μια κορυφαία προτεραιότητα της Ένωσης είναι ότι όταν ε, σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση, ελπίζουμε σύντομα με νέο Πρωθυπουργό, αμέσως να αρχίσει πολιτικός διάλογος και έτσι να γίνουν και τομεακοί αποτελεσματικοί διάλογοι στους τομείς που ενδιαφέρουν. Όπως είπε και ο κύριος Σαφχάουζερ, νομίζω μίλησε για διάγνωση των εξωτερικών δυνάμεων ή κάτι τέτοιο. Κάποια μέλη μίλησαν για τις ρίζες των προβλημάτων. Φυσική πόρη, η εκμετάλλευσή τους είναι ένα τέτοιο θέμα. Προφανώς θέλουμε να δουλέψουμε στα θέματα αυτά ε, ή ε, στην διακίνηση ειδών ε, άγριας πανίδας, αλλά ε, περιοριζόμεθα λίγο γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες διαλόγου και δεν υπάρχει και ε, σχετική ασφάλεια σε σχέση με τους συνομιλητές μας για τον προϋπολογισμό και πώς έχει ετοιμαστεί και πώς ε, τα κονδύλια θα μοιραστούν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Πολλές φορές μας ρωτούν θα υποστηρίξετε τις εκλογές, θα υποστηρίξετε το α, το β και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτή η επιτροπή που πρέπει να συζητήσει το θέμα, αλλά και η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών γιατί έχουμε το θέμα των εκλογών του 2017 και σε ένα εύθραυστο κράτος υπάρχουν πολιτικοί, ε, λειτουργικοί ε, κίνδυνοι, ε, κίνδυνοι πολλών ειδών. Προφανώς βραχυπρόθεσμα έχουμε ηθική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα δεινά του πληθυσμού. Υποστηρίξαμε τον δόκτωρα Μακουέγγιν στο παρελθόν και προφανώς αναγνωρίζουμε τη, μοναδική, τη μοναδικότητα του έργου του. Έχουμε ε, στο Κονγκό και ανθρωπιστική παρουσία και αυτή είναι μια δέσμευση που θα συνεχιστεί. Ούτε μπορούμε να γνωρίσουμε τις ευθύνες που έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Αλλά ουσιαστικά για να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια διαδικασία όπου θα μπορούμε να μιλάμε για μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση, ε, εδώ οι εκλογές είναι το κλειδί και οι πολιτικές διαδικασίες ε, στις οποίες εστιάζουμε τώρα. Κύριε Γκάλερ, νομίζω ότι αναφερθήκατε στο πώς μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά, αν θέλετε, επιτόπου. Προφανώς ε, έχουμε διαδικασίες σχεδίων πήγουσας ανάγκης, αλλά αποφασίσαμε να κλείσουμε τις αποστολές CSTP ε, τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ε, στην ε, μεταρρύθμιση του στρατού παίζουμε ρόλο. Αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρησιακές επιτυχίες. Εδώ θα παίξει ρόλο και το Μονούσκο, αν συνεργάζεται αποτελεσματικά με το SDRDC και θέλουμε να είναι σωστή η εντολή και σωστή η απαραίτητη πόρη που θα τη συνοδεύουν. Ε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανθρώπινη πραγματικότητα ε, στο Ανατολικό Κονγκό ε, η πραγματικότητα ε, σε σχέση με τα δεινά του λαού εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό θα αντιμετωπιστεί κυρίως με αποτελεσματικό κρατικό έλεγχο, ε, με νόμιμες αρχές που θα λογοδοτούν στο λαό. Το τελευταίο που θέλω να πω κυρία Πρόεδρε γιατί μου φαίνεται ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Το τελευταίο λοιπόν που ήθελα να πω αφορά την ευρύτερη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μοναδικός παίκτη που προσπαθεί να πείσει τους πολιτικούς στο Κονγκό να κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση. Συνεργαζόμεθα με την Τανζανία, την Αγγόλα, την Νότια Αφρική, την Ουγγάντα και άλλους παίκτες και την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ. Ε, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις όλους τους βουλευτές και οπωσδήποτε θα τις λάβουμε υπόψη και θα τις προωθήσουμε εκεί που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τους φακέλους του Μπενίν στην κυρία ε, που το ρώτησε. Ε, θα το θέσω στους συντονιστές. μαζί με την, ε, που θα το κάνουν ε, μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σταματήσουμε τις συζητήσεις μας τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, και να σας ζητήσω να κατέβετε κάτω. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 10.30 τώρα. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη γενικά. Uh, outside of hemicycle. Έξω από το ημικύκλιο, στην πλατεία θα συναντηθούμε. Colleagues, please be seated. Thank you. Um, it is my pleasure to... Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά να κηρύξω και πάλι την έναρξη των εργασιών μας μετά την ε, εκδήλωση την τήρηση ενός λεπτού σιγής που είχαμε πριν λίγο μπροστά από το την Ολομέλεια, την αίθουσα της Ολομέλειας. Θα συζητήσουμε το επόμενο σημείο τη ημέρα τη διάταξη, ε, την ε, πολιτική ασφαλείας και άμυνας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και τις επιπτώσεις που έχει αυτή για την Ευρώπη. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές μας, τον κύριο Λέσσερ, Το αντικείμενο της συζήτησής μας όπως είπα, είναι οι πολιτικές ασφαλές και άμυνας των Ηνωμένων και οι πτώσεις που θα έχουν ε, αυτές τις πολιτικές ε, για την Ευρώπη. Καλωσορίζω λοιπόν τους ομιλητές. Ο κύριος Ιαν Λέσσερ, αν, ε, αντιπρόεδρος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ. αρμόδιους θέματα εξωτερική πολιτικής, όπως σας είπα. Ο δεύτερος ομιλητής, ο κ. Στίβεν Μπλόκμανς, από την CEPS. που εργάζεται στις Βρυξέλλες. Και τέλος, ο Γιάνν Γιόελ Άντερσον, αναλυτής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μελετών Ασφαλείας από το Παρίσι. είναι διάρκεια αυτής της συζήτησης θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις απόψεις των ειδικών για τα ζητήματα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα θέμα το οποίο επιθυμούσαμε να συζητήσουμε εδώ και καιρό, ε, μιας και έχουν υπάρξει νέες εξελίξεις μετά τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, συνάδελφοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάντα είχε και συνεχίζει να έχει στενέ σχέσεις με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν θέλετε και για χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, σημαντικές ε, διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά είμαστε και σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έχουμε κάποιες προσδοκίες λοιπόν από τις Ηνωμένε Πολιτείε οι οποίες δράζονται στην ιστορία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έλα πρώτα για κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις και μετά στους ομιλητές. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, διοργανώνουμε από κοινού αυτή τη συζήτηση και θα έχω τη δυνατότητα να συμπροεδρεύσω ω υπεύθυνο και για την ε, ε, ομάδα του Κοινοβουλίου για τη σχέση με τι ΗΠΑ. Γνωρίζουμε ότι, θα, ότι έχουν υπάρξει εξελίξει στα διάφορα κράτη-μέλη με τη μείωση των προπολογισμών για την άμυνα αλλά και στον τομέα του συντονισμού. παρά το γεγονό ότι έχουν υπάρξει περικοπέ και παρά το γεγονό ότι προσπαθούμε να αξιοποιούμε πιο αποτελεσματικά τα χρήματα σε ορισμένου άλλου τομεί πολιτική, θα πρέπει να συνεχιστεί η αποτελεσματική ε, παρουσία τη Ευρώπη, η αποτελεσματική άμυνα και ασφάλεια. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε και την πολιτική κατάσταση. Επισκέφθηκα πρόσφατα την Ουάσιγκτον και από την πλευρά των ΗΠΑ η νέα κυβέρνηση φαίνεται να μετακινείται λίγο από τις θέσεις που είχε εκφράσει προεκλογικά όσον αφορά τις ε, σχέσεις της ε, και τις συμμαχίες της και ε, με το ΝΑΤΟ και να προκινείται προς κάποια μηνύματα τα οποία είναι πιο καθυσυχαστικά, τα οποία εκφράστηκαν και στην πρόσφατη ε, συνάντηση του Πρόεδρου των Πολιτειών με την καγκελάριο Μέρκελ. Ε, ωστόσο παραμένουν πολλά ανοιχτά θέματα και για ορισμένα ε, σκρίσιμες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουν ακόμα διοριστεί από την κυβέρνηση Τραμπ οι αρμόδιοι Σύντομα επίση η, κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει τι ε, ε, θέσεις της για τον νέο προπολογισμό για το 2018. Ε, α, αναμένεται μια αύξηση του προπολογισμού για την άμυνα κατά τη τάξη των 600 εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ακριβώ πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Θα πρέπει ε, επίση να συζητήσουμε με ορισμένα μέλη τη κυβέρνηση των ΗΠΑ της νέας, ε, το ζήτημα τη ρητορική, η οποία μερικέ φορέ μπορεί να δημιουργήσει δυσμενεί επιπτώσει στι σχέσει ε, με. Ευχαριστώ κύριε Έλερ. Τώρα ο κύριο Ιαν Λέσσερ έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σας μιλήσω για αυτά τα θέματα εγώ είμαι Αμερικανός που ζει στις Βρυξέλλες και έτσι έχω μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Συχνά επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον και ο οργανισμός μου είναι Αμερικανικός. Οπότε έχω ένα πόδι και κύθεν του Ατλαντικού και παρακολουθώ του σύνεγγι στα θέματα. Κάτι που απορρέει από αυτά που ακούσαμε τώρα Υπάρχουν κάποιες σημαντικές ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με τις κατευθύνσεις της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ε, διότι, μεταξύ άλλων, πολλοί πολιτικοί που χαράζουν ε, τις πολιτικές δεν έχουν ακόμα καν αναλάβει τα αξιώματά τους. Ε, συνεχίζεται η διαδικασία. Προφανώς υπάρχει μια δομή επαγγελματισμού που τα στηρίζει όλα αυτά και εξασφαλίζει μια συνέχεια. Όμως, οι θέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή η ε, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί κλπ. Ε, οπότε δύσκολα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα και γι' αυτό υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση με τις κατευθύνσεις της πολιτικής και υπάρχει και μια ένταση και μια διαφορά μεταξύ ρητορίας αυτών που λέχθηκαν προεκλογικά και κάποιες ε, διαρθρωτικές δεσμεύσεις από την άλλη. Τρεις παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, πιστεύω ότι η αμερικανική δέσμευση, η βασική και θεμελιώδης για την ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι δομημένη, ανθεκτική, στηρίζεται σε πολλά συμφέροντα και οικονομικά και συμφέροντα κοινωνίας των πολιτών, και αυτά δεν θα αλλάξουν έστω και αν αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Πέρα από αυτά όμως, αν δούμε τις πρακτικές δεσμεύσεις και το γενικότερο κλίμα των σχέσεων, ε, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και θα έλεγα ότι η ιστορική δέσμευση ε, των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα ε, είναι λιγότερο αυτόματες από ό,τι ήταν στο παρελθόν και θα υπάρξουν τριβές εκεί. Το θέμα του επιμερισμού του φορτίου, ποιος πληρώνει τι δηλαδή, δεν είναι καινούριο. Πολλές αμερικανικές κυβερνήσεις ε, έθεσαν το θέμα, πολλές φορές αρκετά αιχμηρά. Οπότε δεν είναι καινούριο που δεν είναι. Αυτό που είναι καινούριο θεωρώ εγώ και θα πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσει να υπάρχει είναι ότι αυτό είναι κομμάτι μιας διαπραγμάτευσης ενεργού. Δεν είναι το θέμα δηλαδή μόνο αν δίνεις αυτά που πρέπει. Σε κάποιες, ε, από κάποιες ομιλίες βλέπω ότι είναι μια διαπραγμάτευση, ένα παζάρι. Δηλαδή, ε, αν δεν πληρώνεις για την άμυνα, δεν θα έχεις άμυνα. Αυτό λένε οι Αμερικανοί και αυτό διαφοροποιείται από την εξωτερική πολιτική της Αμερικής εδώ και χρόνια και την ιστορία των σχέσεων. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό διαπραγμάτευση. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον επιμερισμό των βαρών, αλλά στην Ευρώπη εμείς έχουμε αναλάβει δέσμευση ευρωπαϊκής ασφάλειας γιατί ε, μας ενδιαφέρει, έχουμε συμφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν κάνουμε χάρη δηλαδή σε κανένα, έχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και νομίζω ότι το βασικό, η λιδία λήθος θα είναι αν... ε, ε αυτό ε, συνεχιστεί. Και εκεί υπάρχει η διαφορά μεταξύ των λόγων του Προέδρου και του, των λόγων του άμε, κάποιων από το άμεσο περιβάλλον του και του κατεστημένου γενικότερα. Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σε σχέση με τις ΗΠΑ και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όπως αρέσκονται να λέγουν οι Αμερικανοί. Γιατί εμείς συμμετείχαμε στο εγχείρημα αυτό το σχέδιο Μάρσαλ, έχουμε και το επέτειό του, ο οργανισμός μου ε, έχει ενταχθεί σε αυτή την ιστορία, είμαστε μέρος της, είμαστε βασικοί παίκτες, εμπλεκόμενοι και ε, πολλοί βέβαια στις προηγούμενες δεκαετίες αμφισβήτησαν ε, το θέμα της Ευρώπης και ανταγωνισμού μεταξύ της και του ΝΑΤΟ Πάντα όμως στη βάση ήταν η ιδέα ότι μια πιο συνεκτική Ευρώπη, πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη ήταν ε, υπέρ των Αμερικανικών συμφερόντων. Έτσι θεώρησε το Αμερικανικό κατεστημένο τα θέματα αυτά και οι διαφωνίες ήταν οριακές μέχρι πρόσφατα. Και το αφήνω αυτό ως ανοιχτό ερώτημα. Νομίζω ότι εξακολουθούμε να έχουμε συμφέροντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ε, αυτά θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθούν στο κατεστημένο. Δεύτερον, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική δέσμευση υπέρ της ευρωπαϊκής ασφάλειας εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι σημαντική, υπάρχουν πολλές μεταβλητές εδώ που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ένα είναι η σχέση με τη Ρωσία σε στρατηγικό επίπεδο. Και εκεί δεν θα υπέθετα ότι ε, εκεί κινούμεθα προς ε, μια χρυσή εποχή. Αν δούμε δηλαδή που ταυτίζονται, που διαφοροποιούνται τα συμφέροντα ε, ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας εξαιρουμένης, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Και ο, οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν όταν συναντηθούν, δεν είμαι βέβαιος ότι θα τα πάνε τόσο καλά ε, σε ό,τι αφορά την άμυνα, πυρηνικό εξυγχρονισμό κλπ. Δεν ξέρω. Ε, μάλλον θα είναι τεταμένες οι σχέσεις. Ε, πιο τεταμένες από ό,τι τώρα. Οπότε εδώ αυτό θα παίξει ρόλο υπέρ της συνέχισης της ε, δέσμευσης υπέρ της Ευρώπης. Το, η τρομοκρατία είναι πολύ σημαντικό θέμα, τονίστηκε πάρα πολύ, διέπει όλη τους τη σκέψη και αυτό έχει επιπτώσεις για την άμυνα της Ευρώπης από πλευράς ΙΠΑ. Είμαστε η πλέον στενή εταίρη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σε πολλούς τομείς. Εδώ θα μπορούσα να φανταστώ ε, μια μεσογειακή ε, εταιρική σχέση για την ασφάλεια που αναβαθμίζεται περισσότερο από ότι η σχέση στον κόλφο. Μπορεί δηλαδή να αναβαθμιστεί η Μεσόγειος, να υποβαθμιστεί ο κόλπος. Ε, αυτά είναι κάποιε κάποιες δυναμικές που υπάρχουν που θα επηρεάσουν και τις σχέσεις με την Ευρώπη. Ε, Κορέα, πιο μακροπρόθεσμα η Κίνα, η Ιαπωνία θα μπουν στην ατζέντα της Αμερικανικής ε, κυβέρνησης και θα επηρεάσουν προφανώς και τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Υπάρχουν και ειδικέ εταιρικέ σχέσεις, Τουρκία, δεν θα πω πολλά εδώ, ίσως αργότερα. Ε, μπορεί να είναι σημαντική αλλά δύσκολη η σχέση αυτή. Οι Τούρκοι με κάποια αισιοδοξία τη νέα κυβέρνηση. Μπορεί να είναι πιο ήπιοι σε θέματα ελευθερίας κλπ. Αλλά μπορεί να είναι σκληροί πολύ σκληρή όταν πρόκειται για αιτήματα ε, στα πλαίσια της συνεργασίας για την ασφάλεια. Τέλος, κάποιες νέες προκλήσεις ε, όταν πρόκειται για εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας ε, της νέας διακυβέρνησης είναι καινούρια λόγω ύφους, τόνου, αλλά αν θέλετε οι απαρχές της αλλαγής ε, ανάγονται στο τέλος της διακυβέρνησης Ομπάμα, ο οποίος έκανε πολύ οξύες ε, παρατηρήσεις σε σχέση με την ε, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αν δούμε την συνέντευξή του στο Atlantic Monthly, βλέπετε ότι ο κύριος Ομπάμα είχε γίνει πολύ επιφυλακτικός σε σχέση με την σοφία του κατεστημένου της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, εις ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και θέματα επεμβάσεων. Τέλος, Νομίζω ότι ό,τι και να προτείνει η Αμερικανική κυβέρνηση σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες, ε, την διαφορά μεταξύ ε, ήπιας και σκληρής δύναμης, όλα αυτά θα είναι αντικείμενο διαμόρφωσης από το Κογκρέσο. Θα επηρεαστούν. Και βλέπουμε, ακούμε και από το Κογκρέσο φωνές και από τους στρατιωτικούς φωνές πολύ επικριτικές σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών ε, την, ε, ε, την υποστήριξη για την ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι μπορούμε να περικόψουμε δαπάνες στην ήπια δύναμη, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται εξοπλισμοί. Και νομίζω ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό. Και Τελική παρατήρηση. Πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν για τον απομονωτισμό των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό νομίζω. Ο κίνδυνος, έτσι όπως βλέπετε από τη, μέσα από το πρίσμα των Βρυξελών, έχει, ε, ε, ε, δεν θα είναι τόσο σημαντικός εις ό,τι αφορά πολλούς τομείς συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ο κύριος Στίβεν Μπλόκμαντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε, Πρόεδρε, στην συζήτηση αυτή. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας για την αμερικανική αμυντική πολιτική. Ακόμα λιγότερο μπορώ να ψυχαναλύσω τους Αμερικανούς ε, και το τι θα συμβεί ε, στο μυαλό του, του Τραμπ και στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Αλλά νομίζω ότι κανένας δεν είναι σε αυτόν τον τομέα. Θα περιοριστώ σε τρει παρατηρήσει και δεν θα ε, επαναλάβω. Καταρχάς, υπόθηκαν κάποια πράγματα για τις αμυντικέ δαπάνε από τον συνάδελφο. Συμφωνώ απόλυτα. Η αλλαγή των θεσμικών ισορροπιών εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης. Το υπενήχθηκε ο προλαλή σα. Ένας συνάδελφος, μάλιστα, μας είπε ότι θα είναι η πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού στι ΗΠΑ. Πρώτη στην ιστορία τη. Με τα δικαιώματα των, του Ρεπομπλικανικού κόμματο. ε, από τη μία και από την άλλη ε, ο τραμπισμός. Ε, δεν ξέρουμε ποιος θα πριτανεύσει, ε, ποιος θα κερδίσει. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών ζουν ένα ρήγμα, ένα διχασμό. Ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του ένα σκληρό ισχυρό ηγέτη, περιβάλλεται από τέτοιου ανθρώπου, θέλει να αποδυναμώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Τίλερσον μοιάζει να είναι απομονωμένο ε, από τη γραφειοκρατία, από τη διοίκηση δηλαδή, του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήθελε καν το, την, το φόκο του Υπουργού, αλλά να η γυναίκα του από ό,τι φαίνεται να τον πάρει. Ε, δεν ξέρει όμω τι υποστήριξη καθόλου θα μπορέσει να έχει από τη διοίκησή του, από του υπαλλήλου του, ε, για να μην κάνει περιτά λάθη στη διαδικασία. Ε, Παραδείγματο χάρη δεν πήρε δημοσιογράφου μαζί του στο αυτό το ταξίδι στην Ασία, α πούμε ε, ακούγεται ότι ο Τίλερσον τελικά μπορεί να μην πάει καν στην πρώτη ε, υπουργική, του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο, κάτι που θα στείλει ένα φρικτό μήνυμα στην Ευρώπη. Σε να λέει, α πούμε, ε, πρώτα η Ευρώπη και μετά εσεί. Ε, συγγνώμη, πρώτα η Ρωσία και μετά εσείς Ευρώπη. Από την άλλη έχουμε το Υπουργείο Άμυνα ε, με τον στρατηγό Μάτη, ο οποίο εμπιστεύεται πολύ και δίνει μεγάλη εξουσία και έχει μεγάλη εξουσία. είναι βετεράνος, έχει 40 χρόνια πείρας μέσα σε κυβερνήσεις ξέρει πολύ καλά από πού θα αντλήσει ε, δύναμη. Έχει έμπιστους εκεί, είναι πολύ πιο αποτελεσματικός εντός του Υπουργείου από τον Τίλερσον. Παρότι πολλές ηγετικές θέσεις και στο Υπουργείο Άμυνας ε, παραμένουν κενές. Ε, αυτό μπορεί να τον ε, σπρώξει να αναλάβει, να έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητε και πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Βλέπουμε λοιπόν αλλαγή τη ισορροπία εντό τη κυβέρνηση προς την άμυνα, μακριά από το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το Υπουργείο Άμυνα. Αυτό για την Ευρώπη τι σημαίνει. Ε, το αντίστροφο ε, θέμα, το αντίστροφο ας πούμε ζήτημα, συγκειρικό ζήτημα ας πούμε. Με ποιον θα μιλήσουμε ας πούμε εμείς στην Ευρώπη. Και με ποιον μπορούν να μιλήσουν οι εκπρόσωποι του, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ας πούμε. Μπορούν να μιλήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Ή θα πρέπει να γίνονται δημερώσεις οι επαφές, ας πούμε, από κράτος μέλος, δηλαδή προς την Αμερική κτλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, ε, και το υπενήχθηκε και αυτό η Ιαν, ε, η Αμερικανική πολιτική για την ασφάλεια. Έχουν, το δυναμικό να έρθουν σε αντίφαση ε, και σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές. Πολλοί μιλάνε για το τέλος της στρατηγικής υπομονής ας πούμε, που έκαναν ε, οι Αμερικανοί ε, προς, τη βόρειο, προς την Βόρειο Κορέα. Ίσως πάντως υπάρχει η στρατηγική σχέση με την Νότιο Κορέα, με την Ιαπωνία, κυρίως σε εμπορικά θέματα, αλλά είναι πολύ σημαντική εταίρη σε παγκόσμιο επίπεδο. το πυρηνικό Ιράν. Το πυρηνικό τα πυρηνικά θέματα μάλλον, και, τα, το Ιράν. Πέρα από την, το πώς ξεφυσάει ο Τραμπ, ε, μάλλον θα παραμείνει σταθερό στην πορεία, ε, θα σταθερεί στην πορεία οι Αμερικανοί και θα σεβαστούν, ας πούμε, τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν, για το Συρία, Ιράκ, Μέση Ανατολή. Ο συνασπισμό υπό του Αμερικανού, που υποστηρίζεται από πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον θα παραμείνει δεν βλέπω προς το παρόν μεγάλες διαφορές. Ε, για τη Συρία όμως, ε, το μέλλον του Μπασάρα Λασάντ και η αμερικανική πολιτική μοιάζουν να είναι λίγο ε, στον αδύρα, ας πούμε. Δεν ξέρουμε αν και, η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι σε σύγκρουση. Έχουμε τους Κούρδους, την Τουρκία. Υπάρχει δυναμικός μερίγματος εδώ. Ο μεγάλος άγνωστος χ όμως είναι η Ρωσία. Συμφωνώ με τον Ιαν που πιστεύει ότι δεν θα γίνει μεγάλη αντιστροφή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία, αλλά ίσως υπάρχουν α, κάποιες βυθομετρήσεις, ας πούμε, να τσεκάρουν, ας πούμε, τους ε, Ρώσους Μετά από χρόνια έχουμε, είδαμε ότι 3.500 ε, και μία ε, μεραρχία πέρασε από τη Γερμανία προς την Πολωνία και αναπτύχθηκε στην ε, Βαλτική, Βουλγαρία και Ρουμανία. Τι γίνεται με τα Βαλκάνια. Μόνο με την Ρουμανία που είναι κοντά στη Βουλγαρία ασχολείται προς το παρόν η Αμερική. Δεν νομίζω ότι στα Βαλκάνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη, ειδικά στην Μακεδονία, ούτε καν στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπου έχει μια στρατιωτική αποστολή, στρατιωτική επιχείρηση να για την Ουκρανία και το δυναμικό που υπάρχει. Υπάρχει άμεση επίπτωση της αλλαγής της αμερικανικής πολιτικής ή της αίσθησης της αλλαγής ε, της αμερικανικής πολιτικής ε, στην Ουκρανία και στην προώθηση ας πούμε, της δημοκρατίας ε, παντού σε όλο τον κόσμο αλλά κυρίως στην Ουκρανία. Ε, από την... Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν, υπάρχουν όλα τα, τα συστατικά εδώ, η συμφωνία σύνδεσης, οι κυρώσεις προς την Ρωσία κτλ θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατρανώσει σε επισκέψεις στην Ουάσιγκτον τις θέσεις της και δεν αρκεί η επίσκεψη του Μάικλ. Ε, η προβλεψιμότητα της ε, κυβέρνησης Τραμπ. Λόγω της μια όλο και πιο αυταρχικής Τουρκίας θα πρέπει να αναγκάσει τους Ευρωπαίους να προωθούν σε μια αμυντική ένωση. Υπήρξε έτσι μια, ένα διάλειμμα στην ένταση, αλλά δεν αρκεί αυτό. Επιβεβαιώνει την ιδέα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι μπερδεμένη, ασυνεπείς οι πολιτικές, ε, αυτή η αίσθηση υπάρχει στην Ευρώπη. Ε, η αναξιοπιστία των Αμερικανών προστίθεται στην ε, πολυμερή κρίση της Ευρώπης και θα αποτελέσει τον καταλήτη για μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενδυναμώσουν την συνεργασία για την άμυνα και την ασφάλεια. Ε, αυτό συνδέεται και με το άρθρο 5, το οποίο δεν το κινητοποίησε η Γαλλία. Ζήτησε την ρήτρα αμοιβαία συνεργασία σε άρθρο 42 παράγραφος 7. Ε, αλλά αυτό είναι το προηγούμενο, ας πούμε, για να δουλέψουμε εκτός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ΚΕΠΑ και τη μόνιμη ε, διαρθρωμένη συνεργασία, ε, καθώς και τη δήλωση της Ρώμης, όπου σε τρεις μέρες μπορεί να διατρανωθεί η πιθανότητα για μια, ε, για μια ενισχυμένη συνεργασία στον, στον τομέα αυτό. Ο Ιαν μίλησε για κάποια αδιανόητα μέχρι τώρα. Ε, πυρηνικός πόλεμος, ας πούμε, με τη Βόρεια Εντάξει, δεν το είπες, ε, είναι το αδιανόητο. Τι, πού, τι θέση έχει η Αμερικανή Ε, πόλεμος, ας πούμε, της Κίνας στην θάλασσα της Νότιας Κίνας και απαγγελία κατηγορίας εναντίον του, του Τραμπ. Ε, ή να το αφήσουμε να κυλήσει γιατί αποκλείεται να συμβούν όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γιάννη Ιωελ Άντερσον. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι ιδιαίτερο ευτυχή για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που θα έχω να συζητήσουμε. Οι θέσεις που θα αναπτύξω είναι προσωπικές, ε, γιατί για τα θέματα αυτά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Μελετών ε, Ασφαλείας δεν έχει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Είναι δική μου ανάλυση λοιπόν. Σημερίζομαι την αίσθηση των προλαλήσαντων, αλλά έχω και κάποιες διαφορετικές ε, αξιολογήσεις. Και έχω προετοιμάσει επίσης και μια ε, παρουσίαση με διαφάνειες, γιατί έχω διαπιστώσει τη σημασία που έχει το να χρησιμοποιεί κανείς διαφάνειες από τις παρουσιάσεις που έχω κάνει σε στρατιωτικούς κάθε το παρελθόν. Εν ολίγης, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει συνέχεια, όχι μόνο στη ρητορική, αλλά και στην πολιτική. Μακροπρόθεσμα, όμως, και είναι ζήτημα ορισμού ότι είναι μακροπρόθεσμο και την είναι πρόθεσμο. ε, ίσως υπάρχουν αλλαγές. Και αυτό, σε αυτά αναφέρθηκε και κανείς και συνάδελφοι. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι συνυπάρχει μια ρητορική η οποία εκφράζεται στο υψηλότερο επίπεδο, στο επίπεδο του Πρόεδρου, για παράδειγμα, και ε, η καθημερινή διαχείριση που γίνεται. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού θα οδηγηθούν οι σχέσεις των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ, οι διμερείς τους σχέσεις με κράτη της Ευρώπης εξαιτίας αυτής της ρητορική. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την προεκλογική ρητορική. Αυτή ήταν ε, αυστηρή και επικριτική προς την Ευρώπη. Και πολλοί Αμερικανοί από think tank, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρθηκαν στα ζητήματα του, ε, του του οικονομικού κόστου τη άμυνα τη Ευρώπη, αλλά αυτό είναι για εσωτερική κατανάλωση, πιστεύω. Ότι μας λένε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για αυτό. Όμω αυτό που ανταπαντούσαμε είναι ότι ναι, αλλά αυτά είναι σε δημοσιοθέα, τα ακούει όλο ο κόσμο. Άρα ακόμα και αν λέγονται για εσωτερική κατανάλωση στις ΗΠΑ, Πολιτείες, υπάρχουν επιπτώσεις γιατί ακούγονται διεθνώς. Ο, ο πρόεδρος Τραμπ συνέχισε να εκφράζεται με τρόπο παρόμοιο με εκείνο που είχε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Και παρόμοιες θέσεις έχουν εκφραστεί τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό Άμυνα. και συνεχίζει να μας προβληματίζει αυτή η ένταση και αυτή η διαφοροποίηση μάλλον που υπάρχει μεταξύ του Προέδρου και υψηλόβαθμων υπουργό του ή ακόμα και του Αντιπροέδρου. Αυτό έχει περιγραφεί ε, και εξηγηθεί αν θέλετε από το γεγονό ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν τρία-τέσσερα επίπεδα λήψη αποφάσεων. Φανταστείτε Πώ λειτουργούν τα πράγματα στις δικέ σας ε, χώρε, που φυσικά δεν υπάρχουν τρία-τέσσερα επίπεδα, αλλά η μετάβαση του μήνυματο από πάνω προ τα κάτω παίρνει χρόνο. Και το συμπέρασμα είναι ότι για του επόμενου 6 με 8 μήνε δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή. Θετικό είναι αυτό, αλλά και πάλι μιλάμε για το βραχυπρόθεσμο. Βραχυπρόθεσμα πάντως δεν πρέπει να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Ένα άλλο λόγο που δεν περιμένουμε μεγάλε αλλαγέ βραχυπροθέσμου είναι επειδή οι πολιτικέ οι οποίε αυτή τη στιγμή ακολουθείται δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Για παράδειγμα, η πολιτική ευρωπαϊκών εγγύσεων, στην πρωτοβουλία ευρωπαϊκών εγγύσεων στην Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να υφίσταται από το 2014 και τώρα ε, το 2017 έχει, έχει ε, προγραμματιστεί η μεταβάσεις, η οι αλλαγές των ε, σταθμιμένων ε, στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτείων. Το γεγονό ότι έχουν αναπτυχθεί αμερικανικέ δυνάμει στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη ε, χρειάστηκε μια προετοιμασία δύο-τριών ετών. Έχουν προγραμματιστεί ασκήσει και αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να σταματήσουν. Πρόκειται για ασκήσεις οι οποίες ε, έχουν μεγενθυνθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύσεων. Έχουμε 28 ε, πολυμερείς ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν 18.000 ε, Αμερικανοί στρατιώτες και 45.000 στρατιώτες από χώρες του ΝΑΤΟ. Και αυτό επίσης οδηγεί σε, στην πρακτική συνεργασία των στρατευμάτων ε, επιτόπου. Επομένως το μήνυμα που δίδεται είναι ότι το... οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ε, παρουσία στην Ευρώπη ότι... και, και αυτό ε, έχει σημασία και για Αμερικανούς στρατιωτικούς να συνεχιστεί. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν πρόκειται να αλλάξει ο διοικητή ούτε τη ε, USEUCOM ούτε τη SACUR, τη ανώτατη συμμαχική διοίκηση. Επομένω, Και τέλο υπάρχει και οι σχέσει και η υποστήριξη που έχουν στο Κογκρέσο αυτέ οι επιχειρήσει. Όμως, για τι εξελίξει μακροπρόθεσμα, πέρα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ο Ιωάννη και ο Στίβεν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ορισμένες από, τις, από τους όρους που έχουν ακουστεί, από τις φράσεις που έχουν ακουστεί. Να βάλουμε την Αμερική πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Οι φράσεις αυτές δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι σημαίνουν στην πράξη. Και παρόλο που ακούγονται εντυπωσιακέ και ισχυρέ, είναι ε, αμφίσιμες. Μπορεί να ερμηνευτούν από πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και ο τρόπος με τον οποίο θα ερμηνευτούν πιστεύω ότι θα έχει επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως για παράδειγμα η σύνδεση με ε, την ε, αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική. κατά πόσον θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της αλλαγής πολιτικής ή ακόμα και να αναπληρώσουμε το κενό. Οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής στην αμερικανική πολιτική θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν σε αυτήν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι θα, αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό οι δαπάνε για την άμυνα θα μπορούσε να έχει επιπτώσει και για την οικονομία γενικότερα και για την προοπτική τη οικονομία. Το 2017 έχουμε διάφορε εκλογικέ ανεμετρήσει στην Ευρώπη που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Και επίση το 2018 με τι εκλογέ για το Κογκρέσο θα δούμε και πώ θα συνεχιστεί πώς, θα ε, εξελιχθούν τα πράγματα στην Ουάσιγκτον και αν τελικά αυτός ο συνασπισμός που περιέγραψε ο Στίβεν θα συνεχιστεί. Ο τρόπος αντιμετώπιση αντιμετώπισης, αυτό για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, είναι αντιμετώπιση κρίσεων. Είτε στη Λιβύη, είτε στι εξελίξεις στην Αφρική, είτε σε πιθανές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, πρέπει να προετοιμαζόμαστε ετοιμαστούμε μακροπρόθεσμα για να έχουμε τη δυνατότητα ανταπόκριση σε κρίσεις. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μερικές φορές οι Αμερικανοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον όρο Multilate ε, Παίζοντα με τις λέξεις εννοώντα ότι είναι μια σειρά πολυμερών σχέσεων με τι Ηνωμένε Πολυεπίπεδη. Ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει από ένα επίπεδο και να περάσει στο επόμενο. Όμως, Υπάρχει μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη σχέση της με τις ΗΠΑ Πολιτείες και είναι μια άλλη συζήτηση του πώς θα εξελιχθεί η σχέση με τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα πάμε προς μια διαφοροποίηση, περισσότερη σύγκληση εκεί. Επίσης δεν θα πρέπει να υποτιμούμε την δυνατότητα, την ικανότητα των Ευρωπαίων να διχάζονται και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στη σχέση με τους Αμερικανούς. Το... Υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την ε, Ουάσιγκτον, την Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία. Υπάρχουν διάφορες χώρες στην Ευρώπη που θεωρούν ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Και οι Αμερικανοί είναι πολύ ικανοί στο να μας ε, τα καταφέρουν καλά, στο να μας κάνουν να το πιστεύουμε αυτό. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρώπη να διχαστεί και πάλι. Όμως υπάρχει και μια ευκαιρία και μια ε, ευθύνη αν θέλετε να το λαμβάνουμε αυτόν υπόψη μας, την πιθανότητα διχασμού δηλαδή και να το προλαβαίνουμε στη σχέση μας με τις ΗΠΑ. αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο του Βιετνάμ ή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα για το Ιράκ. Εγώ θα σταθώ στις γνώσεις που έχω από την σχέση των ΗΠΑ με την Σουηδία, η οποία ήταν πολύ τεταμένη κατά τη διάρκεια της, της περίοδου του πολέμου στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί απέσυραν τον πρέσβη του από τη Στοκχόλμη την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργό τότε ε, εκφραζόταν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Παρόλα αυτά, εκείνη την εποχή, η πολιτική και η στρατηγική συνεργασία συνεχίστηκε χωρίς κανένα πρόβλημα με μεταφορά τεχνογνωσίας, ε, συνεργασία τεχνολογική, πωλήσει όπλων, ανάπτυξη νέων ε, τεχνολογιών κτλ. Το οποίο μας δείχνει ότι η πολιτική και η στρατιωτική συνεργασία, ιδιαίτερα σε τεταμένες περιόδους, αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Φανταστείτε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, των αμερικανικών ε, εταιριών ε, ή των ευρωπαϊκών εταιριών μάλλον που συνεργάζονται ε, και με την αμυντική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή επίσης τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις και τις σχέσεις που υπάρχουν στο επίπεδο το ανώτερο, το, στρα, το, το στρατιωτικό. Αμερικανοί διοικητέ, Αμερικανοί στρατηγοί που επισκέπτονται ε, τους ομολόγους τους στις ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα. Κλείνοντας και προσπαθώντας να κλείσω ένα συμπέρασμα, έχουμε από τη μια την ε, προεκλογική ρητορική και από την άλλη την συνέχεια. Ε, βρισκόμαστε στην αρχή της, της ε, Προεδρίας Τραμπ και θα εξελιχθούν τα πράγματα συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την στην Ευρωπαϊκή Άμυνα θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, αλλά, ε, βράχη πρόθεσμα, συγγνώμη, αλλά μακροπρόθεσμα παραμένουν διάφορα ερωτηματικά. Στο πώ θα εξελιχθεί, για παράδειγμα, η σχέση με το ΝΑΤΟ. Και εμεί, ω Ευρωπαίοι έχουμε επιλογέ στη, στη, στη διάθεσή μας και πρέπει να επιλέξουμε πώ θέλουμε να κινηθούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη περίοδο θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις, πολλά γεγονότα, ε, όλο και πιο πυκνά τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ για την πολύ καλή ενημέρωση από τους τρεις συμμετέχοντες. Φοβούμαι ότι ίσως κάποιοι στην Ευρώπη που βασίζονταν αποκλειστικά στις ΗΠΑ, στις σχέσεις τους και μέσα από το ΝΑΤΟ, νιώθουν σαν την εγκαταλειμμένη νύφη, όπου ο σύζυγος ε, λέει κάποια λέει πλατωνικές υποσχέσεις, εκτός κι αν η νύφη δώσει γερή πρίκα. Και εγώ ε, θέλω να κάνω πολιτική δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος του 2%. Είναι για το δικό μας το συμφέρον, πέρα από αυτό που θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Γιατί εδώ ε, υπάρχει κάποια έγκυρη κριτική, ε, έγκυρη κριτική ότι οι Αμερικανοί το λένε και το είχαν πει και πριν. Ο κύριος Λέσερ είδα ότι αναφέρθηκε στην άποψη των προηγούμενων διακυβερνήσεων ότι η πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική Ευρώπη είναι, ε, για το είναι υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων. Ισχύει αυτό και τώρα, γιατί χρειάζονται ειδικά σε αυτό το στάδιο κοινά σαφή μηνύματα που τώρα πρέπει να πάνε στους παραλήπτες που πρέπει στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή το μήνυμα μέχρι τώρα ήταν σαφές, πιστεύετε. Και είναι πιθανό στην πράξη να δούμε να ασκείται μια πολιτική από το Πεντάγωνο και τον ΙΠΕΞ μαζί με το Κογκρέσο όταν πρόκειται για χρηματοδότηση και ε... ε άμυνα που θα ε... αποκλίνει από το Λευκό Οίκο. Δηλαδή τα καθήλυν ε, αρμόδια υπουργεία μπορεί να κάνουν μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρη για την ε, συνέχεια. Ο κύριος Φρόιντ θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, όχι θέλω. Θέλω και παραθέλω. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Μπλόκμαν που είπε ότι δεν πρέπει να είναι κανείς ψυχολόγος για να αξιολογήσει ε, τα λεγόμενα του κυρίου Τραμπ. Ε, κάποιος πιο ηλικιωμένος από τους περισσότερους εδώ έχει παρακολουθήσει πολλές ε, αμερικανικές κυβερνήσεις για πολλά χρόνια. Ποτέ όμως δεν είδα μετά την αλλαγή από τον Κάρτερ στον Ρέιγαν, από τον Μπούς στον Κλίντον ή από τον Τζορτζ Μπούς στον Μπαράκ Ομπάμα Ποτέ δεν είδα τον πρόεδρο και όχι προεκλογικά, αλλά μετά την εκλογή του δεν έχω ξαναδεί πρόεδρο να κάνει tweet λέγοντας για τον προκάτοχό του ότι είναι άρρωστος, ότι είναι κακός. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα, οπότε δεν πρέπει να είναι κανείς ψυχολόγος για να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Διάβασα στις 2 Ιανουαρίου ένα άρθρο που προέβλεπε κάτι που φαίνεται να γίνεται ότι στις 20 ε, ε, ε, Ιουνίου η Βόρεια Κορέα θα εκτοξεύσει πυράβλους βαλιστικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το, η στρατιωτική... Ε, θα έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους, θα τηλεφωνήσουν μέσα στη νύχτα στον πρόεδρο για να του πούν ότι έχουμε θέμα με την Κορέα. Και λέει με τον Τσικ Κορέα είχατε θέμα. Όχι, με τη Βόρεια Κορέα. Και έρχεται και ακούει τα διάφορα σενάρια που παρουσιάζονται γιατί ε, ο πύραυλος έρχεται και δεν ξέρουν πού θα πέσει στη θάλασσα, στον ειρηνικό ή πιο κοντά στην ακτή. Οπότε η μία ακτη οποτε λέει να κάνουμε το α, η άλλη πλευρά λέει να κάνουμε το β. Και μετά ο, ο πρίμπους νομίζω ε, λέ, είπαν ότι είπαν, ε, κύριε πρόεδρε, στο, στο χέρι σας είναι να αποφασίσετε. Και αυτό είναι που με φοβίζει εμένα, γιατί θα αποφασίσει πάνω σε ποια βάση. Οπότε σας ρωτώ, ε, βαίνομαι προς μία πολύ φρικτή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θα αναφερθώ σε μια παρατήρηση του Ιαν Λέσσερ ότι το θέμα δεν είναι ο αμερικανικός ε, απομονωτισμός, αλλά η αμερικανική μονομέρεια. Οι Αμερικανοί για την Ευρώπη θέλουν έναν ισχυρό αξιόπιστο εταίρο για να μοιράζονται τα βάρη. Είπατε ότι οι ΙΠΑ πάντα υποστήριζαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό ανάγεται στη δεκαετία του 40, τη δεκαετία του 50, πολύ διαφορετικές εποχές όταν ήταν κατεστραμμένη η Ευρώπη και έπρεπε να ξανά επανοικοδομηθεί η οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών και βέβαια υπήρχε και η σοβιετική απειλή τότε και έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να επανεντάξουμε την Γερμανία στην άμυνα των δημοκρατιών μας. Περί αυτού επρόκειτο τότε. Τρόποντινά μπορεί κανείς να πει σχεδόν ότι ξαναπέζεται το ίδιο έργο. Και το ερώτημά μου είναι πώς επανεντάσουμε πάλι τη Γερμανία ώστε να μην ε, ανησυχήσουν οι, ευρωπαϊκοί, οι ευρωπαίοι γείτονες ε, της Ευρώπης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με διπλασιασμό αμυντικών δαπανών, μάλλον απίθανο. Όταν μιλάμε όμως για 2% περί αυτού πρόκειται διπλασιασμό των αμυντικών δαπανών της Γερμανίας. Και ξαναγυρίζουμε στο παλιό ερώτημα. Πώς ε, χειριζόμεθα μια τέτοια ισχυρή Γερμανία πλέον και οικονομικά και στρατιωτικά. Εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί η απάντηση σε αυτό που δεν έχει λεχθεί είναι ότι θα μπορούσε η Γερμανία να ενταχθεί στην ευρύτερη, στο ευρύτερο αυτό μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω λοιπόν να θέσω και Επίσης, ξαναγυρίζω στο θέμα της μονοπλευρης πολιτικής. Αν δούμε τις μονομέρειες, αν δούμε τα παραδείγματα που ανέφερε ο κύριος Άντερσον, που είπε για το Βιετνάμ, υπάρχει και άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα που ε, ανησυχεί τους Ευρωπαίους. η Σύνοδος Κορυφής το 86 μεταξύ Ρέιγκαν και Κορμπατσόφ. Ανησύχησαν τότε οι Ευρωπαίοι γιατί σκέφτηκαν ξαφνικά «Ω Θεέ μου, θα συμφωνήσουν οι δυο τους πάνω από το δικό μας το κεφάλι, θα στερήσουν την Ευρώπη από την πυρηνική ομπρέλα που τη θέλαμε για να αποτρέψουμε συμβατικούς πολέμους ε, στην Ευρώπη». Αυτό ήταν μια ανησυχία. Και αν θυμάστε, ε, αυτό ήταν και το κίνητρο, ανοήτως κατ' να ε, αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να γίνει μια προσπάθεια να ε, υπάρξει η ιδέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευρωπαϊκή ικανότητα. Το έθεσα αυτό γιατί τα παραδείγματα της μονομέρειας των ΙΠΑ είχαν καλοήθης αν θέλετε επιπτώσεις γιατί αν δούμε τι έγινε μετά τη Σύνοδο Κορυφής του 86 οδήγησε σε μείωση εξοπλισμών αλλά και στη μετέπειτα κατάρρευση της ε, Σοβιετικής Ένωσης και όλα όσα έγιναν μετά. Δεν είμαι βέβαιος ότι πρέπει να ανησυχούμε ε, οπωσδήποτε, αλλά με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας σχετικά με το ποιες μορφές μπορεί να πάρει αυτή η μονομερής πολιτική και τι συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί. Και ξαναγυρίζω ότι οι ΙΠΑ χρειάζονται ε, ισχυρούς και αξιόπιστους εταίρους. Και το πρόβλημα στο οποίο επανέρχομαι και είναι παλιό σχετικά με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, αμυντικές της φιλοδοξίες, γιατί πέρα από, πέρα από και από το γερμανικό ζήτημα, το πρόβλημα νομίζω είναι ότι αυτοί που μιλούν για την ευρωπαϊκή άμυνα, δηλαδή την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, δεν ε, οδηγεί σε αυξημένη στρατιωτική ικανότητα, ενώ μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια υπηρετική Ευρώπη που θα είναι λιγότερο αξιόπιστη ως εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργηθεί μια επιρωτική Ευρώπη, η οποία αν θέλετε έχει στρατηγικές φιλοδοξίες δικές της, θεωρώντας αυτήν ως διαφορετικό παράγοντο, παράγοντα ε, παγκοσμίω, χωριστά από τις ΗΠΑ. Και δεν ξέρω αν είναι τόσο μικρός ο κόσμος ώστε να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί από μόνη της. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει η συμμαχική σχέση και τι είναι αυτά που μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ και τι δεν μπορεί να κάνει. Όχι να εφεύρουμε πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ, αλλά να δούμε τι όντω δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ και πού μπορούν να παρέμβουν άλλοι οργανισμοί οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορέσουν να συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι ε, δεν θέλω να ε, μιλάμε ε, εντελώ θεωρητικά για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ, ας πούμε ενδεχόμενος ρόλος του στην Αφρική, ότι είπα δεν έχουν συμφέροντα εκεί κλπ. Θα πρέπει να δούμε τι όντως δεν μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ, ποιος δεν είναι ο ρόλος του. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις δικές μου και ε, θα ήθελα τη γνώμη και των ε, ειδικών μας. Κύριε Βαλέρο. Thank you. I, um, I have a question... Μία ερώτηση. Να ξεκινήσω καταρχάς λέγοντας ότι είμαστε όλοι κατάπληκτοι με τις δηλώσεις Τραμπ ε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Παρότι ήταν για εσωτερική κατανάλωση, συνεχίζει να λέει τις ίδιες ακρότητες. Όταν τον ακούγαμε κατά διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είχα την αίσθηση ότι αν γινόταν πρόεδρος, θα τον σταματήσουν. Όταν προσγειωθεί στην πραγματικότητα, όταν αναλάβει τη θέση του ως πρόεδρος, ε, υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες, διάφορα επίπεδα, τα οποία θα πρέπει να σεβαστείς, όπως είπε και ο Ιαν, και ότι θα τον ελέγξουν δεν μπορεί να κάνει, ότι θα μπορούσε να εγκλωπίσει όλα όσα έλεγε. Όμως τίθεται το ερώτημα, μια και είσαστε κι εσείς πολιτικοί, ξέρετε ότι έχουμε ιδέες, έχεις ιδέες ως πολιτικός, τις λες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, μετά γίνεσαι μέρος του συστήματος και σε σταματάνε. Αλλά όχι για πολύ, γιατί μπορεί να αλλάξει τους κανόνες επειδή είσαι μέρος του συστήματος. Και το ενδιαφέρον είναι τι γίνεται μακροπρόθεσμα. Κύριε Γλέσσερ, μακροπρόθεσμα, πώς βλέπετε τα πράγματα, ποιες είναι οι προοπτικές του Τραμπ, τι δυνατότητες έχει για να υλοποιήσει αυτά που είπε ότι θέλει να κάνει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει κάποιες ιδέες, θέλει να τις αναπτύξει, θέλει να, ήθελε να κλείσει τα σύνορα ας πούμε. Βρήκε κάποια προβλήματα που τον ανέκοψαν, αλλά τελικά προχωράει. Μακροπρόθεσμα τελικά τι θα γίνει όμως, τι θα μπορέσει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Μπλόκμαν. Θα ήθελα να μιλήσετε περισσότερο για αυτή την ξεχασμένη θέση που είναι, έχει βρεθεί η Συρία και το θέμα των Κούρδων κτλ. Και εγώ νομίζω ότι η Συρία έχει πέσει σε αυτή την ε, ξεχασμένη θέση. Ποιος Πολύ ενδιαφέρουσα τα σχόλια. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λέσσερ και άλλοι ομιλητέ. Ότι πρέπει να απομακρυνθούμε λιγάκι από τον τύπο, από τη μορφή που πήρε η συζήτηση, μέσα από τις δηλώσεις, μέσα από τις ρητορίες του Τραμπ. Είναι ρητορίες οι οποίες μας σοκάρουν, μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να έχουμε πολλές αβεβαιότητες. Πίσω όμως από τον τύπο υπάρχουν ουσιαστικές τάσεις στο εσωτερικό της Αμερικανικής κυβέρνησης και στρατηγικές τάσεις επίσης αμερικανικές που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, τόσο άρδιν. Πολύ σωστό είναι αυτό που είπατε, ότι τα αμερικανικά αιτήματα από τους Ευρωπαίους εταίρους είναι πανάρχαια. Απλώς εκφράζονται διαφορετικά. Παλιότερα εκφράζονταν πιο ευγενικά. Θυμάμαι την ε, συζήτηση του και το λόγο του κύριου Γκέιτς εδώ στις Βρυξέλλες πριν από έξι χρόνια ήταν αρκετό ομός θα έλεγα τότε. Θυμηθείτε την ε, κυβέρνηση Κλίντον η οποία ήταν ε, μια κυβέρνηση που λάτρευαν οι Ευρωπαίοι η οποία όμως δεν ήταν πάρα πολύ συμφιλωτική και δεν συνέκλεινε με τις προσπάθειες που κάνουν οι Ευρωπαίοι να οργανωθούν μόνοι τους. Μην ξεχνάτε τι είχε πει Όλμπράιτ για τις τάσεις της αμυντική Ευρώπη τη Ευρώπη που προωθεί τη δική τη άμυνα. Αυτέ οι τάσει των Αμερικανών υπάρχουν εδώ και χρόνια και υπενθυμίζουν στου Ευρωπαίους τι ευθύνε του. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, Απλώ τα, τα λέει διαφορετικά τώρα ο Τραμπ και πολύ πιο σοκαριστικά, αλλά η ουσία δεν έχει αλλάξει άρδιν. Για αυτή την ιστορία του 2%, αυτό το, το θέμα, α πούμε, του 2% ΑΕΠ. Εγώ ανήκω σε μια χώρα επιτρέψτε να μιλήσω λιγάκι ψαγάλο, ή μεγάλος, που δεν φτάνει στο 2%. Αλλά ποιο θα αμφισβητήσει, σα παρακαλώ, τι στρατιωτικέ προσπάθειε που κάνει η Γαλλία. Για ελάτε να μου πείτε. Γιατί και μονομερό και διμερό και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη δεν βλέπω πολλέ άλλε χώρε που κάνουν όσα κάνει η Γαλλία. Το ίδιο και στι επενδύσει, στι αμυντικέ επενδύσει. Επενδύσει δηλαδή σε αμυντικού εξοπλισμού. Το 2% εντάξει, καλό είναι, ένα στόχο. Μπορούμε να, προσπαθήσουμε να τον υλοποιήσουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτά. Γιατί μπορεί να έχει ένα τεράστιο προπολογισμό αμυντικό, αν δεν κάνει τίποτα με αυτό, τι νόημα έχει να τον έχει. Επομένω, προσοχή, προσοχή. Μην κολλάμε πάρα πολύ σε τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Ε, τώρα, λίγο προκλητικά θα ήθελα να πω ότι αν έχετε απλώ 1% ας πούμε, του ΑΕΠ που το δίνετε στην άμυνα, αλλά με αυτό το 1% ε, έχετε εξοπλισμούς, αγοράζετε τα πάντα από τους Αμερικανούς, σε αυτά που σας ε, ε, προτείνουν ας πούμε προς πώληση, προφανώς θα τους αρέσει, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους αρέσει ακόμη και αν είναι το 1%. Επομένως να τα δούμε όλα αυτά έτσι μέσα στο σωστό πλαίσιο. Μετά από αυτό το σχόλιο, μία ερώτηση για την Αφρική, που είναι ο ξεχασμένο παράγοντα ε, σε αυτέ τι συζητήσει και τι παρουσιάσει. Και είναι ένα θέατρο παρόλα αυτά, όπου και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί είναι πολύ δραστήριοι και συχνά μαζί. Μέσω δύο αξώνων τριών μάλλον. Καταρχάς, τις ε, αμερικανικές ε, δράσεις, 100% αμερικανικές. Οι Αμερικανοί έχουν στρατιωτικέ επιχειρήσεις σημαντικές, παρότι είναι διακριτικές στην Αφρική. Παραδείγματος χάρη, στο κέρα τη Αφρικής, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται ε, στη Σομαλία, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν επί προεδρία Ομπάμα, τι θα γίνει με αυτή τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση. Θα αμφισβητηθεί, θα εντατικοποιηθεί, θα μείνει στο ίδιο επίπεδο, τι θα γίνει. Υπάρχουν επίσης οι μικτές, δρά... οι μικτές προσπάθειες. Ε, οι, παραδείγματος χάρη, Αμερικανοί που στηρίζουν τις ε, γαλλικές προσπάθειες ε, στο Σαχέλ, ας πούμε, που είναι διακριτική η βοήθεια, αλλά είναι ουσιαστική. Ε, ειδικές δυνάμεις, αεροπορική στήριξη, είναι σημαντική η αμερικανική αυτή βοήθεια. Είναι ένας από τους άγνωστους χι της ε, νέα κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε να γίνεται λόγο. Αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί ε, των Αμερικανών ενώ, ή θα μπορούσαν να το θυσιάσουν οι Αμερικανοί αυτό. Και τρίτο ερώτημα, ε, το τρίτο είδος δέσμευση και παρέμβασης στην ε, Αφρική, που είναι λιγάκι άχρωμο και άοσμο, γιατί δεν έχει τη φραγίδα των Αμερικανών είναι μέσω του ΟΗΕ, ας πούμε, και τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Ο πρόεδρο ε, όμω ε, διέταξε μια αναθεώρηση ε, εντελώ δραστική των Αμερικανικών προσπαθειών και τη δεσμευσή του απέναντι στο ΟΗΕ. Και δεν αγγίζει μόνο τι ήπιε δράσει, ας πούμε, αλλά και τι ειρηνευτικέ, που είναι πάρα πολλέ, πολύ σημαντικέ και χωρί κατάλληλη χρηματοδότηση μπορούν να καταρρεύσουν. Και οι Αφρικανικέ χώρε, οι οποίε αποφελήθηκαν θα διαλυθούν περαιτέρω. Αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Τι πιστεύετε για αυτή την αναθεώρηση που διέταξε ο Τραμπ ε, αυτών των δραστηριοτήτων πούμε, και των παρεμβάσεων που κάνει ο ΟΗΕ στην Αφρική. Ο κ. Ανδρουλάκης, παρακαλώ. I'm very sorry. Ε, ο κ. Ντροιεύσκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσα και ενδελεχής η ανάλυση. Λοιπόν, η πολιτική άμυνας δεν δέχεται κενά. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη, ε, ένας αντίπαλος μπορεί το κενό να το αξιοποιήσει υπέρ αυτού. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ανάλυση μάκρο και βράχη πρόθεσμη. Το κενό ε, αρμοδιοτήτων θα πρέπει να εξεταστεί στα δύο αυτά επίπεδα. Υπάρχει ε, πρόβλημα στην Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει επίσης ένταση του, μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας. Η οικονομική αλλά και η πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία επιδεινώνεται. Ε, πολλοί πολλές συλλήψεις έγιναν και ε, το Σάββατο κλιμακώθηκε η κρίση στο Μίνσκα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει απειλή στην περιοχή. Ε, ε, υπάρχουν στρατιωτικοί ε, χειρισμοί που προβλέπονται στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν αυτά τα πρωτόγνωρα γεγονότα. Επίσης έχουμε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και εκεί υπάρχουν εντάσεις. Στη Γεωργία επίσης τα προγνωστικά δεν είναι καλά. Πρέπει λοιπόν οι παρατηρητές, οι αναλυτές να φροντίσουν να ασκηθούν πιέσεις, ούτως ώστε το κενό αυτό αρμοδιότητας να πληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Στην περίπτωση της Κρυμαίας ε, μας ξεπέρασαν οι εξελίξεις, παρόλο που είχαμε έγκαιρες προειδοποιήσεις για τις εξελίξεις στην Κρυμαία. Κι όμως δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες, να τις αναλύσουμε και να τις σταθμίσουμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να προβλέψουμε το κακό και να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στις ε, ε, σαφώς διαφαινόμενες απειλές. Ε, Επίση στην Ουκρανία η κατάσταση είναι αποσταθεροποιημένη. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία και υπάρχουν και πολλές απειλές που και αυτές μπορούν να ε, οδηγήσουν σε σοβαρές ε, συνέπειες όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και για όλη την Ευρώπη. Με ενδιαφέρει το εξή. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε μόνο έναν απολογισμό, να κάνουμε μια ανάλυση και να εκείνο που πρέπει είναι να αντλήσουμε συμπεράσματα ε, μαζί με τους Αμερικανούς, ούτως ώστε το κενό ε, αρμοδιότητας να πληρωθεί. Σημαντική είναι και η οικονομική παρέμβαση από το... και η παρέμβαση από το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε μήπως ε, υπάρχουν λάθος τάσεις, υπάρχουν ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε και σε επίπεδο ανάλυσης και σε επίπεδο οικονομικής υποστήριξης για να αντιμετωπίσουμε ε, τις μεγάλες απειλές που παρατηρούμε στην Ενδοτική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που προκύπτει για μένα ξεκάθαρα είναι ότι είναι ένας άγνωστος χ η αμερικανική πολιτική για όλους σχεδόν. Το μόνο απτό και πραγματικό είναι η γεωστρατηγική ε, μετακίνηση των Αμερικανών προς την Ασία και υποβάθμιση της σχέσης της Ευρώπης για τους Αμερικανούς. Από την άλλη, ε, η επιμονή για αυτό το 2%. Ευτυχώς, ε, μετά από τις έντονες δηλώσεις για την Ταϊβάν, ε, υπήρξε μία έτσι αποκλιμάκωση και ελπίζω να επιβεβαιωθεί σε επόμενες συνεδριάσεις με την Κίνα. Εμείς θα θέλαμε όλη αυτή η νέα στάση να οδηγήσει σε μια ανεξάρτητη βεβαίως ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντιβαίνει στο ΝΑΤΟ. Όχι. Χρειαζόμαστε μια αυτόνομη πολιτική, αμυντική πολιτική. Δεν νομίζουμε ότι είναι λάθος το να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική αμυντική και πολιτική ασφάλειας και ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με, την, με τον ΝΑΤΟ. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Μεσόγειο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, μια προσπάθεια προς τη δική μας γειτονία. Θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπε η συνάδελφος Βαλέρο για το ρόλο των Κούρδων στη Συρία. Ε, υπάρχουν τρεις βάσεις ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, η Ρωσία όμως άνοιξε ότι θα ανοίξει και μία νέα βάση στο Κουρδιστάν της Συρίας. μπορεί να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία ε, μεταξύ Αμερικανών Ρώσων για την ε, Συρία. Ε, η Ευρώπη είναι εκτός των συζητήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι κακό, κακή είδηση. Ε, εκεί που γίνονται σημαντικές εξελίξεις ας πούμε, και σημαντικές αλλαγές σε στρατιωτικό επίπεδο ε, είναι λάθος να απέχουμε. Ούτε στην Γενέβη βρισκόμαστε. Ε, Ε, αν βάζουμε ας πούμε κυρώσεις και δεν μιλάμε καν ας πούμε με τον έναν από τους δύο εταίρους μας ας πούμε ε, νομίζω ότι θα γυρίσει αυτό που μένει βάρος μας. Και μια άλλη ερώτηση για το Ιράν. Πιστεύετε ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική για το μη πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων ε, για το στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σχέλος. Χθες ο Ιρανός Υπουργός ε, άμυνας, υπεύθυνο για, σημαντικά ε, για σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις, είπε ότι δεν πρόκειται μέχρι, έτσι, μέσω πρόθεσμα να φτιάξουν ε, πυρηνικά όπλα στο Ιράν. Εκτός από τους τακτικούς πυράβλους που έχουν να κάνουν με την ε, άμυνα τους απέναντι στο Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικό το Ιράν ε, για το ρόλο που μπορεί να παίξει στον άξονα εκεί της Μέσης Ανατολής ε, και για τη Συρία. Αυτά ευχαριστώ. Thank you now, Mr. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνεται την αδυναμία ε, της Αμερικανικής Γερουσίας εξαιτίας της άρνησης του Ρεπουμπλικάνου Γερουσιαστή Ραντ Πολ την προηγούμενη εβδομάδα να εγκριθεί συμφωνία ένταξης του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ. Και δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς πιστεύετε ότι θα συμπεριφερθεί η πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς θα αντιμετωπίσει την ε, κατάσταση στην Τουρκία με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μετά το δημοψήφισμα θα γίνει ένας απόλυτος άρχοντας, θα πάμε σε μια μορφή εσωτερικής απολυταρχίας, όπου σίγουρα θα, δημιουργεί, θα εντάσεις και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά σύνορα της Τουρκίας. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση του κύριου Τραμπ και της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ, που έφυγα, αλλά μου, είπαν τι διεμήχθη στο μεταξύ. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση και να μιλήσω λιγάκι για την πολιτική του Τραμπ. Την βρίσκω διαφανή, ξεκάθαρη, πεντακάθαρη. Αντίθετα από όλα όσα ακούγονται για αυτήν. Καταρχάς, η αρχή της ευθύνης και της ε, προ, πρωταρχικής σημασίας των αμερικανικών συμφερόντων. Κάθε κράτο, α πούμε, περασπίζει με υπεύθυνο τρόπο τα συμφέροντά του. Είναι κλασική αρχή τη διπλωματίας και χτίζει συμμαχίε με βάση τα συμφέροντά του. Προτιμώ χίλιε φορέ αυτή την πολιτική από την ε, πολιτική της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, ε, και όπου στην πραγματικότητα ε, στην πραγματικότητα η Αμερική χρησιμοποιώντας ας πούμε χρησιμοποιούσε τη Συρία, τη Λιβύη, ε, τις διάφορες επαναστάσεις στην Αραβική κτλ. Έπαιζε ένα πολύ άσχημο ρόλο, αλλά είχε κάθε υποτίθεται ηθική ας πούμε, δικαιολογία. Ενώ εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική, η οποία υπερασπίζει τα δικά της συμφέροντα. Με ισορροπημένο τρόπο προσπαθεί να βρει συμμάχους τέλεια, τέλεια. Να μια πραγματική πολιτική η οποία δεν ε, αιματοκυλάει τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά, αυτό τι σημαίνει, ότι εμείς από την πλευρά μας αναλαμβάνουμε τις ευρωπαϊκές μας ευθύνες. Μιλήσαμε για τις ευθύνες της Γαλλίας, το είπε ο συνάδελφος. Η Γαλλία, κατά την άποψή μου, ήταν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ θέλουμε να βγούμε από το ΝΑΤΟ, αλλά καταλαβαίνω ότι οι χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να συμμετέχουν οικονομικά. Λογικό είναι. Τουλάχιστον καταβάλουν το 2% του ΑΕΠ τους για τις αμυντικές ανάγκες του ΝΑΤΟ. Ένας υπουργός οικονομικών, Γάλλος, είπε ότι αν η Γερμανία είχε ξοδέψει τα ίδια ποσά με τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, μετά τον πόλεμο δηλαδή, αλλά ξέρω δεν το έκανε, έτσι, τότε το χρέος της Γαλλίας θα ήταν το ίδιο με της Γερμανίας. Θα είμαστε δηλαδή σε μία πολύ πιο άνετη θέση οικονομική, αν δεν το είχαμε κάνει ας πούμε. Είναι, είναι νούμερα τα οποία τα είπε ένας δεξιός υπουργό ε, οικονομικών, έτσι, συμμαχός σας. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μαζί με τα μέλη του, Υπουργείου του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, να συνεργαστούμε. Ε, αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι απόλυτα διαφανές. Θέλει μαζί με αυτούς να φτιάξει μια παγκόσμια ε, συμμαχία, πούμε, και μια ισορροπία ε, που θα είναι ικανή να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Εσύ, εσείς που είσαστε ε, η παλιά φρουρά του Κλίντον, δεν βλέπετε ας πούμε αυτό το New Deal της Αμερικής, γιατί είσαστε μέσα στα ιδεολογήματά σας κολλημένοι. Εγώ που είμαι ανοιχτό, που δεν είμαι ανταμερικανός, ε, που ήμουνα μαζί σα όταν θέλετε να καταπολεμήσουμε τον κομμουνισμό. Το βρίσκω λοιπόν τέλειο αυτό που κάνει ο Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι ευκαιρία για την Ευρώπη και αν τη χάσουμε θα είναι δράμα. Σα ευχαριστώ. Thank you. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και κύριε Έλερ, σας δίνω το λόγο με οποιαδήποτε ιδιότητα θέλετε, είτε αντιπρόεδρος της ΕΔΕ, είτε άλλη ιδιότητα που έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μιλήσω ως Γερμανός αρχικά. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας αφενός και μεταξύ Γερμανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά η Γερμανία έχει πολλές υποχρεώσεις, επίσης έναντι του ΝΑΤΟ. Και, Τζέφρι, ε, χαίρομαι για τις ευφύς αναλύσεις σας, αλλά βλέπουμε τους τόρις στο Ηνωμένο Βασίλειο να πηγαίνουν από τον 20ο αιώνα και πίσω πίσω πίσω στο 19ο, δεν ξέρω πια που θα οδηγήσει αυτό. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Το ζήτημα δεν είναι πλέον πώς θα προστατεύσουμε την Ευρώπη από τη Γερμανία. Αναμφίβολα, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες. Όμως ρωτώ τους ειδικού. από τα 660 εκατομμύρια αύξηση του, του αμερικανικού προϋπολογισμού, αυτό που αναλογεί στην Ευρώπη είναι 30 εκατομμύρια. Ε, γιατί οι υπολογισμοί που κάνουν οι Αμερικανοί για την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών δεν σχετίζονται άμεσα με τον ΝΑΤΟ. Και όπως είπε και ο κ. Φανόρντεν, εάν αύξηναν οι δαπιντικές δαπάνες στα 62 δι, το ερώτημα τελικά θα τεθεί για να τα κάνουμε τι, για να, για να, για να τα αξιοποιήσουμε πώς αυτό σχετίζεται με το στρατηγικό ρόλο του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να ανταποκριθεί στην, στο ρόλο που του τον παραδοσιακό, ως συμμαχία δηλαδή, ή περιμένουμε από το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει και ζητήματα όπως η τρομοκρατία, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, όπως η κατάρρευση κρατών. Το ερώτημα που γεννάται. Γιατί είναι κάτι που θα συζητηθεί, ε, συζητήθηκε στην Ήτρε και συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αυτή η δημιουργία ενός ε, μια συμμαχία σε μεσογειακό επίπεδο, στο οποίο θα συμμετείχαν και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, με προγράμματα αναπτυξιακά ανάπτυξης και έρευνας στον τομέα της άμυνας, αλλά φυσικά και περαιτέρω συνεργασία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι επιδιώκουμε ως μείγμα πολιτικής είναι αύξηση των εξοπλισμών, των παραδοσιακών, είναι δαπάνες περισσότερο για τομείς ασφάλειας τους οποίους έχουμε παραμελήσει ή αυτό που λέγεται να να αυξήσουν χώρε όπω η Γαλλία, η Γερμανία και άλλε τέτοιε μεγάλε χώρε του προπολογισμού του για να φτάσουν στο 2% του ΑΕΠ. Βεβαίω όλα αυτά μετρώνται σχετικά με το ΑΕΠ. Και αν δει κανεί το ποσοστό των αμυντικών δαπανών τη Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ τη είναι πολύ μεγάλο. Αν μιλάμε για το ΑΕΠ μια χώρας όπως η Γερμανία, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αναλογικά το ποσοστό είναι μικρότερο. Το ερώτημα λοιπόν που θέτω είναι ε, εμεί, εσεί τι περιμένουμε να υιοθετήσουμε ω μείγμα πολιτικής άμυνα και εξωτερικών. Και πιο πρακτικά, τι περιμένουμε από το ΝΑΤΟ τον, στον τομέα τη καταπολέμησης της τρομοκρατίας εάν υπάρξει το ενδεχόμενο να υπάρξει μπλοκάρισμα από την πλευρά της Τουρκίας των, των πρωτοβουλειών εντός του ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μια άλλη ένα άλλο κέντρο, ε, άλλη διοίκηση αν η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να συνενέσει. ή αναλλακτικά θα, περίμενε κανείς μια μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ τώρα ως απλό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που έκανε ο κύριος Έλερ Και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχω βαθιά πίστη στους ελέγχους και στην ισορροπία τη θεσμική του Αμερικανικού συστήματος. Το οποίο με οδηγεί σε κάποιες σκέψεις. Θα ήθελα να ξανασκεφτούμε λίγο αυτά που τον κύριο Ντονζάν και ο κύριο Στρογεύσκη. Απ' τη μια έχουμε πολλές προκλήσεις της όσον αφορά την παγκόσμια ασφάλεια παντού στον κόσμο και από την άλλη έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες που έχουν τη δυνατότητα να μας ε, υποστηρίζουν ακόμα και, σε ένα περίπλοκο πολιτικό ε, τοπίο. Υπάρχουν πολλοί τομεί συνεργασία και πολλοί τομεί του οποίου συνεισφέρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και οποτεδήποτε αποσύρονται οι Αμερικανοί, δημιουργείται ένα κενό το οποίο οδηγεί σε συγκρούσεις και περαιτέρω προβλήματα. Άρα είναι απαραίτητο να βρούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό επιδιώκουμε ε, ταυτόχρονα να ε, αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ, ταυτό, ενώ ταυτόχρονα είναι δύσκολο να καταλήγουμε σε συνελετικές λύσεις. Δύσκολα συμφωνούμε στην ανάλυση μας για το ποιες είναι οι απειλές. Άρα χρειάζεται κατά την απόψη μου περισσότερη σε συντονισμός περισσότερη ενοποίηση στον τομέα της ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας για να καταλήξουμε σε μια κοινή αντίληψη για το ποιε είναι οι απειλές που ε, αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και έρχομαι σε αυτό που είπα. Στην... Όπως πιστεύω ότι είναι αποτελεσματική η θεσμική ισορροπία και ε, η έλεγχη πολυεπίπεδη στην Αμερική, Ταυτόχρονα με ανησυχεί η τρέχουσα κατάσταση. Είναι λιγάκι διαφορετικό το θέμα, αλλά σχετίζεται και με όλα τα ζητήματα που συζητάμε ως τώρα. Αυτό που με ανησυχεί λοιπόν είναι η κατάσταση του προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και το ότι θα χρειαστεί να ληφθούν αποφάσεις εξισορρόπηση διαφορετικών τομέων πολιτικής, διαφορετικών δαπανών. Και κάτι ακόμα που αφορά περισσότερο τη δικιά μα Ήπειρο, είναι η, η ε, χρήση του, το στάτους του δολαρίου ως ε, το νόμισμα που χρήσει η παγκόσμια οικονομία. Και εδώ πρέπει να δούμε εάν ε, είμαστε ε, συνεκτικοί εμείς ως κράτη-μέλη της Ευρώπης και αν ε, υποστηρίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν υποστηρίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να έχουν προκεχωρημένη παρουσία και να επεμβαίνουν για την προστασία και για την σταθεροποίηση ε, γεωγραφικών περιοχών στις οποίες έχουμε από κοινού συμφέρον να είναι σταθερές. ίσως να μην είναι εδώ το κατάλληλο φόρουμ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά σίγουρα οι κύριοι έχουν αλλάξει, έχουμε ένα πόλεμο πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα. Και παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα της άσκησης της αμερικανικής πολιτικής. Εγώ θα έλεγα ότι ε, είμαι περισσότερο ήσυχη. Γιατί φαντάζομαι ότι βραχυπρόθεσμα ή και μέσο πρόθεσμα δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Βεβαίω, όσον αφορά το τι θα συμβεί στι πολιτικέ μακροπρόθεσμα, είναι πιο άγνωστο, είναι λιγότερο γνωστό, αλλά εδώ που τα λέμε, κανεί δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον μακροπρόθεσμα. Άρα κανένας από εμά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει τόσο συνεκτικές πολιτικές που να τις έχει σχεδιάσει πλήρως ως το μέλλον. Ε, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς στην Πολωνία και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το αναφέρω και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το τι συμβαίνει στις φυλακές στη Συρία. που πλέον επιβεβαιώνεται από τη μαρτυρία εκείνου που κατάφερε να φύγει από τη Συρία και να φέρει φωτογραφίες που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου σε μαζική κλίμακα στις φυλακές. η συνάντηση των συμμάχων στην Ουάσιγκτον. Στην συνάντηση αυτή συμμετέχουν χώρες οι οποίες υποστηρίζουν τον Ασάντ ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Το ερώτημα λοιπόν που έχω εγώ είναι πώς θα βρούμε έναν κοινό παρονομαστή τις πολιτικές μας επιδιώξεις. έτσι ώστε να συντονιστούμε εν ώψη και του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές του πάνελ με την ίδια σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που βάλατε Πολύ ενδιαφέροντα όλα βέβαια. Δεν θα τα σχολιάσω όλα. Πολλοί μίλησαν για τον πρόεδρο Τραμπ και πώς ενδέχεται να απαντήσει σε μια κρίση. Βέβαια, οι εικασίες σχετικά με τη συμπεριφορά μιας κυβέρνησης σε σταθερή κατάσταση είναι ένα θέμα και το άλλο Άλλο είναι να προσπαθήσεις να βολιδοσκοπήσεις πώς θα αντιδράσεις σε μεγάλη κρίση ασφάλειας ή οικονομική κρίση. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του ανδρός αλλά και με τη δυναμική ε, του στο Λευκό Οίκο και ε, αλλού. Είναι ε, κρίσιμο το ερώτημα. Δεύτερον, αυτό που είπε ο Τζέφρι Βαν σχετικά με την πιο συνεκτική ε, Ευρώπη και πιο συνεκτική και πα... Συνεκτική είναι. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο του κύριο Βαν Δεν ήταν. Όχι, γιατί συζητούνται αυτά και στις ΗΠΑ. υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα, κάποιες ανησυχίες. Πάντως, ε, διαχρονικά, οι ΙΠΑ καθησύχασαν σε σχέση με την Ευρώπη για διάφορους λόγους. Δεν ανησυχούν τόσο πολύ για τον ανταγωνισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Άμυνας. Σωστό ή λάθος. Πάντως, σωστό είναι να πούμε ότι η βασική άποψη της Washington άλλαξε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πιο άνετη τώρα σε σχέση με όλα αυτά. Τώρα, η, αυτή η κυβέρνηση διαφοροποιείται. Ε, δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούν τα ίδια ε, μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει κανείς για να ε, τους πείσει είναι να πάει και να τους πει στην Washington ότι αυτός ο τρόπος έχει καλή σχέση κόστους ωφέλειας και καλό θα ήταν να υποστηριχθεί η λύση αυτή αν δεν θέλουμε κατακαιρματισμένο Ευρωπαίο εταίρο αλλά πιο συνεκτικό, θα πρέπει να συμφωνήσετε με την πρόταση. Μπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ερώτημα για τη Γερμανία. Κέριο ζήτημα προφανώς και είναι κρίσιμο να δούμε την ουσία της πρόσφατης συνάντησης Μέρκελ-Τραμπ. Υπάρχουν φωνές στην κυβέρνηση αυτή που επικρίνουν πολύ τη Γερμανία σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο για την άμυνα αλλά και την εμπορική πολιτική και άλλα πολλά. Και θα ανησυχούσα γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι βασικό συμφέρον για είπα να έχει εταίρο τη Γερμανία και αντίστροφα. Από άποψη εμπορική δηλαδή. Ναι, καλό θα ήταν να ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα που είχε αρχίσει και ήθελε να ολοκληρώσει ο Ομπάμα, το, η συμφωνία TTIP και όλα τα συναφή ναι, που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν είναι καλό για την αμυντική συνεργασία να γίνεται μάχη για την θεωρητικά καλή πολιτική ε, εμπορίου ε, εργασίας κλπ. Ε, ε, πολλοί λένε δεν πρέπει να ανησυχούμε για την Κίνα αλλά για τη Γερμανία. Αυτό είναι μια σημαντική μετακίνηση στο τοπίο της Ουάσιγκτον. Τώρα, αν θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένη πρακτική αλλαγή πολιτικής δεν ξέρω. Αυτό πάει χέρι με χέρι με την επιδείνωση, όπως έδεισε ο Πολ, στην ε, γερμανική κοινή γνώμη. Αυτό το, το έδειξαν οι δημοσκοπήσεις, θέλω να πω διατλαντικές σχέσεις εξαρτώνται ε, από τη στάση του, του εκάστοτε ε, Αμερικανού Προέδρου. Οπότε αυτά τα θέματα έχουν σημασία. Υπήρχε 60% εμπιστοσύνη στις ε, ΗΠΑ παλιότερα και τώρα έπεσε στο 20% και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις η πτώση είναι πολύ στατιστικά πολύ σημαντική. Εγώ περιγράφω την κατάσταση ως έχει και το θέμα του τριπλού μηδέν και όλα αυτά είναι σωστά. Η, αυτή η μονομέρεια, η προβληματική, τι μορφή μπορεί να πάρει για την Ευρώπη. Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα εδώ. Τώρα μπορεί να πάρει τη μορφή ότι θα δραστηριοποιηθούν στην άμεση γειτονία της Ευρώπης η ΗΠΑ χωρίς να διαβουλευθούν ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ ή να συναποφασίσουν για τις στρατηγικές, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Σίγουρα ε, η Ευρώπη παίζει ρόλο για την σταθερότητα σε σχέση με τη ε, Ρωσία που ενδιαφέρει τις ΕΠΑ. αν ε, υπάρξει ε, νέος ανταγωνισμός εξοπλισμών, πυρηνικών εξοπλισμών, δεν θα προκύψει τίποτα, ούτε θα μειωθεί ο κίνδυνος. Ό,τι κάνουν οι ΙΠΑ σε αυτό το μέτωπο θα ενδιαφέρει την Ευρώπη, είτε τη διαβουλευτούν είτε όχι. Ε, το θέμα της Αφρικής είναι πολύ σημαντικό. Ή ΙΠΑ ΕΕ νομίζω ότι θα εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στην Αφρική με, στα πλαίσια της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας. Και είναι αλήθεια ότι αν δούμε ποια χώρα στην Ευρώπη ήταν η πιο ε, δραστήρια σε αυτό το τομέα, ήταν η Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια λέω. Οπότε και αυτό είναι μια άλλη κρίσιμη διάσταση των σχέσεων μεταξύ υπάρχει και Ευρώπη. Τώρα, πού δαπανώνται τα κονδύλια. Είναι σημαντικό αυτό και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί ο πρόεδρος λέει να ψηθούν οι δαπάνες, αλλά αυτό που θα ενδιαφέρει τα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η αντιμετώπιση χαοτικών καταστάσεων. Ε, αυτό δε, όμως δεν είναι αυτό που στοιχίζει, δεν είναι τόσο δαπανηρή η διαδικασία αυτή. αυτο δε ομως δεν ειναι αυτο που στοιχιζει δεν ειναι τοσο δαπανηρη η διαδικασια αυτη πολλά δαπανώνται στο, στο μέτωπο εσωτερική ασφάλειας, πολιτική εκεί. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό μεταξύ των ετοιμάτων των ΙΠΑ και του μεγάλου ενδιαφέροντο που έχει, δηλαδή την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και εκεί ο οικονομικός παράγον δεν είναι τόσο σημαντικός. Ε, τώρα, τώρα, ε, ΙΠΑ, Τουρκία, σίγουρα ξεχνώ πολλά. Για την Τουρκία είναι πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το αν θα γίνει καλύτερη η σχέση. Πάντα περιγράφεται ως στρατηγική η σχέση ΙΠΑ-Τουρκίας, αλλά πάντα δύσκολα αντιμετωπίζονταν για διάφορους λόγους. Πολλές φορές ε, χώρες δραστηριοποιούνται καθαρά για ίδιο συμφέρον. Δύο πράγματα θέλει η Τουρκία από τη ΣΥΠΑ. Θέλει ε, να απελαθούν και να εκδοθούν ορισμένοι θεωρούμενοι αντίπαλοι και να αντιμετωπιστούν το θέμα ε, των εμπόλεμων στη Συρία. Θα είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιήσει τα δύο αυτά αιτήματα η παρούσα κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη για παρόμοιους λόγους. Υπάρχουν ε, διαδικασίες στα δικαστήρια για τον Γιουλέν, θα πρέπει να περιμένουμε τι θα γίνει. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους Τούρκους. Για το κουρδικό και τις δυνάμεις των Κούρδων στη Συρία, αυτή η κυβέρνηση ε, θα λάβει μάλλον σκληρότερα μέτρα εις ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και το ποιος βοηθάει και ποιος όχι. Οι Κούρδοι θα πρέπει να αξιολογηθούν πάνω σε αυτή τη βάση. Ε, θα είναι δύσκολο οι Τούρκοι να πείσουν τους Αμερικανούς να μην συνεργάζονται με τους Κούρδους. Τέλος, αν μπορώ να σχολιάσω και να απαντήσω στην ερώτηση για τα εθνικά συμφέροντα εναντί άλλων ε, παραμέτρων. Προφανώς τα εθνικά συμφέροντα ε, καλό είναι να ε, προάγονται, ε, ιδιαίτερα για μια παγκόσμια δύναμη. Αλλά αυτό είναι περιορισμένο η άποψή μου είναι, όχι της κυβέρνησης, αναγκαστικά, ότι ε, έχουμε ένα συστημικό συμφέρον να μην εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση ο κόσμος, δηλαδή να προάγει μόνο εθνικά συμφέροντα. Εύκολα μπορεί να υπάρξουν ανταγωνισμοί και να κλιμακωθούν αυτοί και μπορεί να ξαναγυρίσουμε στη δεκαετία του 30. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε μια τέτοια εμπειρία. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που θέλουμε, δεν θα είναι σταθερός ε, μπορεί να ε, έχουμε κάποια αιτήματα βάσει εθνικής κυριαρχίας, αλλά αυτά δεν ε, μπορούν να συγκεράζονται με την ανάγκη για μια παγκόσμια τάξη. Ευχαριστώ. Κύριος Μπλόκμαντς, ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις. Πάρα πολλές, θα σταθώ σε λίγες. Και να έρθω σε αντίφαση ε, μάλλον να διαψεύσω αυτά που είπε ο Ιαν για την Τουρκία, έτσι για να παίξω το δικηγόρο του διαβόλου. Να ξεκινήσω ε, με το, το σχόλιο του Τζέφρι Βαν Όρντεν για την ε, ενίσχυση του ΝΑΤΟ, που είναι πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο. Αν και την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ασφάλεια και την άμυνα, για να δούμε πού μπορούμε να δράσουμε συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ. την περασμένη εβδομάδα στην Εστονία είδα ότι η Εστονία βασίζεται στο ΝΑΤΟ και σε τάγματα και άρματα μάχης ε, υπό την αιγύδα των Αμερικανών που, που έχουν αναπτυχθεί εκεί. Ε, θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι συμπληρώνει στην κυβερνοάμυνα, στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλύτερη να το κάνει αυτό, αυτό θεωρούν οι Αμερικάνοι, ε, καθώς και στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο ε, που δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εκεί όπου δραστηριοποιείται μπορεί να είναι πολύ πιο σε φάση, ας πούμε, συντονισμένη, ας πούμε, πολύ περισσότερο από ότι το ΝΑΤΟ με κάποιες χώρες κτλ. Ε, τώρα, Τουρκία-ΝΑΤΟ. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξανασκεφτεί τη διαδικασία ένταξης ε, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και δεν σε τα πολιτικά κριτήρια της Κοπενχάγης, ε, παρόλα αυτά πρέπει και το ΝΑΤΟ να το σκεφτεί αυτό το θέμα. Καταρχάς, αξιακά μπορούμε να βασιστούμε σε, έναν, ένα αυταρχικό καθεστώς, αυταρχικό σύμμαχο, αλλά και μετά τα, τις εκαθαρίσεις του μετά το πραξικόπημα χθε ε, πέρυσι, ε, πολλά υπουργεία, πολλές υπηρεσίες, ε, στρατός κτλ. Ε, στην πραγματικότητα διαλύονται και ο Ερντοάν δημιουργεί μια πρετοριανή φρουρά εκτός συστήματος. Μπορεί το ΝΑΤΟ να συνεχίζει να βασίζεται λοιπόν σε ένα τέτοιο σύμμαχο Τουρκία είναι βασικό θέμα, πολιτικά σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προβληματίζεται για τη θέση της απέναντι στην Τουρκία και πώ θα προστατεύσει τα δικά τη δηλαδή στρατηγικά συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Μετά την Τουρκία περνάω στο θέμα των Κούρδων. Συμφωνώ ότι προς το παρόν ε, είμαστε σε, στην ίδια φάση εμείς με τους Αμερικανούς για την υποστήριξη του Κουρδιστάν και το YPG της ε, πολιτοφυλακής ε, κουρδικής ε, Συριακής όπου η Άγκυρα βέβαια πιέζει και, την, και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους να τους στυλιτεύσουν ως τρομοκράτες αυτή την πολιτοφυλακή. Εδώ διαφέρω λιγάκι, διαφωνώ λιγάκι με, τον, με την ανάλυση του Ιαν. Η YPG ήταν αξιόπαστος εταίρος για τους Αμερικανούς ε, πολεμώντας τη Συρία. Παρ' όλα αυτά θα τους πετάξουν οι Αμερικανοί από το παράθυρο όταν γίνει μια ευρύτερη συμφωνία για τη Συρία. Ή δεν θέλουν Ξέρετε πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί μερικέ φορέ δεν υπερασπίζονται του συμμάχου του στην ε, Μέση Ανατολή και δεν καταλαβαίνω. Όταν το YPG, αυτή η πολιτοφυλακή παίξει το ρόλο τη, δεν φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν οι Αμερικανοί να του στηρίζουν. Θα του ξεφορτωθούν. Η Real Politik εδώ θα υποδείξει τα συμφέροντα των Αμερικανών. Και συμφωνώ με αυτού που είπαν ότι υπ' αυτή την έννοια οι πολιτικέ των Αμερικανών, ναι, είναι διαφανεί. Είναι διαφανεί. Όμω συμφωνώ και με κάτι που είπε ο Ιαν, ο Ιαν ότι σε κρίσεις ο ανώτατος διοικητή αποφασίζει και χρειαζόμαστε πραγματικά εδώ ένα ψυχαναλυτή και για τη Βόρεια Κορέα. Δεν υπήρξε κάποια αντίφαση σε κάποιε δηλώσεις νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε ψυχανάλυση του Τραμπ γιατί τα συμφέροντα δεν άλλαξαν τίποτα δεν άλλαξε και ε, ο Λευκός Οίκο πάντα θα παίξει το ρόλο του. Αλλά σε κρίσει εξαρτώμαστε περισσότερο ε, από προσωπικότητες. Ποιο θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει εκείνο ή θα πει στο μάτι εσύ αποφάσισε. Ο Υπουργό Άμυνα. Αυτό είναι σημαντικό. Σα ευχαριστώ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι συνάδελφοι ήδη έχουν απαντήσει σε πολλέ ερωτήσει. Θα ήθελα γι' αυτό να μιλήσω για αυτά που παραμένουν ανοιχτά. Οι εκλογές έχουν επιπτώσεις, υπάρχουν αλλαγές, αλλάζουν την πολιτική, ιδιαίτερα σε ένα προεδρικό σύστημα όπως εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό η εκλογή προέδρου έχει μεγάλες επιπτώσεις. Ε, ακόμα περισσότερο τώρα που υπήρξε και αλλαγή στο Κογκρέσο και στην Γερουσία. Επομένως, Κατά μία έννοια μπορεί κανείς να πει ότι όποιος κερδίσει τις εκλογές έχει και το δικαίωμα να αξιοποιήσει αυτή του τη νίκη. Το γεγονό ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη κατά του διατάγματος του Τραμπ για τους μετανάστες δείχνουν ότι υπάρχουν και θεσμικές, ε, θεσμικοί έλεγχοι ε, αυτό θα εξελιχθεί, αλλά επίσης υπάρχει και το Κογκρέσο, το οποίο ελέγχει τον προϋπολογισμό, ελέγχει τις δαπάνες και όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του Ρεπλουπλικανικού Κόμματος που υποστηρίζει την συνεχιζόμενη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Υπάρχει μια, αν θέλετε, γενιά πολιτικών που έχει γαλουχηθεί ε, ε, ε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και αυτή τη στιγμή φεύγουν σιγά σιγά, ο κύριος Κέιν για παράδειγμα. Και στην κυβέρνηση μπαίνουν νέα πρόσωπα σε εκθέσεις κλειδιά που θα προωθήσουν τις δικές τους απόψεις και κατά την άποψή μου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν κάτι ανάλογο του Κογκρέσου για την Ευρώπη, έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Όσον αφορά τώρα τη σχέση, τη, τη συζήτηση για το ΝΑΤΟ από τη μια ή την μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας. Εδώ ε, δεν υπάρχει πλήρης αλληλοεπικάλυψη των συμφερόντων ή των αρμοδιοτήτων. Των ΝΑΤΟ έχει μια παγκόσμια πολιτική. Την προστασία, για παράδειγμα, ε, μέχρι και των τηλεπικοινωνιακών γραμμών σε ε, ε, απομακρυσμένους ωκεανούς. Αυτά, αυτά είναι θέματα τα οποία θα απασχολούσαν μια δύναμη νατοϊκή ή την ανάπτυξη δυνάμεων σε χώρες τη της Αφρικής. Ε, και υπ' αυτή την έννοια σε τέτοιου τομεί δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των, ενδιαφε... των συμφερόντων και των επιδιώξεων τη Ευρώπη και του ΝΑΤΟ. Τώρα για τη σχέση με την Τουρκία. Ε, συμφωνώ με τι ανησυχίε που εκφράστηκαν. Ήδη αυτή την εβδομάδα ε, τέθη θέμα με το μπλοκάρισμα από την πλευρά της Τουρκίας της συνεργασίες της Αυστρίας με τον ΝΑΤΟ. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει τεταμένη σχέση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. πρέπει να σκεφτούμε και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχουν οι τεταμένες σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Και αυτό είναι ακόμα πιο ενισχυτικό. Πριν δύο χρόνια έγραψα ένα μικρό άρθρο για τις ε, σφιγμομετρήσεις που έγιναν στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, για το κατά πόσον οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θέλουν να υπάρξει άμυνα, να, να, φροντίζει οι, να φροντίζουν οι ΗΠΑ για την άμυνα της Ευρώπης. Και ένα μεγάλο μέρος των ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων ήταν υπέρ της ε, εμπλοκής των ΗΠΑ για να προστατεύσουν την Ευρώπη από την απειλή τη Ρωσική. Όμως, αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να αλλάξει. όπως αναφέρθηκε από τους συνομιλητές, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξουν οι προτεραιότητες όταν πια λέγεται ότι η Γερμανία είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από την Κίνα. Επομένως, έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε σε πιο πεζά θέματα, αν θέλετε, σε πιο απλή και τεχνική συνεργασία, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ. 30, μισό λεπτό. Ε, υπάρχει ανακοίνωση ε, σχετικά ε, με τη συμμετοχή στην ε, συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Έχει επιβεβαιωθεί δηλαδή η συμμετοχή της κυβέρνησής του. Ε, ωραία, ευχαριστώ πολύ όλους. Νομίζω ότι ε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Ε, ελάτε και το απόγευμα γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης η απογευματινή συνεδρίαση. Και ευχαριστώ τη Γραμματεία γιατί μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε συζήτηση ενδιαφέρουσα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Ε, θα με πράγματα που δημιουργούν διλήμματα ασφάλειας, όπως π.χ. Ε, την κατάσταση στην Ανατολική και Νότια Κινέζικη θάλασσα, και θα μιλήσουμε και για την πολιτική ασφάλεια της Ιαπωνίας. Ελάτε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σημειώνω ότι αρχίζουμε στις 3 και 4 το απόγευμα. Ευχαριστώ.